Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Θα αρχίσουμε. Έχουμε διάφορα μικρά πραγματάκια πριν περάσουμε στο κυρίως θέμα μας που είναι η κοινή συζήτηση της Επιτροπής μας Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με κύριο θέμα την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη και πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Πριν περάσουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα ουσία, σας περάσουμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Εδώ υπάρχουν δύο αλλαγές που έχω να σας προτείνω. Η πρώτη είναι ότι προσθέτουμε ένα νέο σημείο 4α που είναι τα πρακτικά των συντονιστών. Και δεύτερον, ο Σεπτάνς που είναι εισηγητής ε, γνωμοδότησης, συντάκτης γνωμοδότησης για τον κατάλογο σίγουρων χωρών, θέλει το δικό του το σημείο αύριο το απόγευμα να περάσει δηλαδή το 23 πριν από το 20. Οπότε το σημείο 23 που είναι το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική θα είναι αύριο γύρω στις 4 και το σημείο 20 που είναι ο Ενωσιακός Κοινός Κατάλογος Ασφαλών Χωρών, θα εξεταστεί στις 6. Ελπίζω να συμφωνείτε με τις τροποποίησεις αυτές. Οι βοηθοί παρακαλώ να ενημερώσουν ε, τους συναδέρφους, τους κοιόδης, για να ξέρουν τι ώρα θα εξεταστεί ποιο σημείο και ανάλογα να έρθουν. Δεύτερο σημείο, ανακοινώσει της Προέδρου. Δεν έχω ανακοινώσει. Αύριο το πρωί στις 9 ψηφίζουμε. Παρακαλώ να είσαστε στην ώρα σας. Ξέρω ότι κλείνει, τώρα το απόγευμα έχει κλείσει η la Λαλουά, οπότε πολύ δύσκολο να φτάσουν οι συνάδελφοι. Σημείο 3. Ανακοινώσει τη Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι έχουμε τίποτα από την ΤΕΦΚΟ, σωστά. Δεν υπάρχουν ανακοινώσει λοιπόν ούτε από την Επιτροπή. Σημείο 4. Έγκριση των πρακτικών. Πρόκειται για τα πρακτικά της συνεδρίασης της 25ης Ιανουαρίου. Είναι στους φακέλους σας. Αν έχετε παρατηρήσεις, να ενημερώσετε την γραμματεία πριν τη λήξη της συνεδρίασης. Αλλιώς, τα πρακτικά θεωρούνται εγκεκριμένα. Σημείο 4α. Έχετε και τις αποφάσεις και συστάσεις των ε, συντονιστών της 17ης Αν έχετε παρατηρήσεις ή οτιδήποτε άλλο, να μας το πείτε. Αλλιώς θεωρούνται εγκεκριμένα και αυτά τα πρακτικά των συντονιστών. Οπότε, αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα περνάμε στο κυρίως θέμα μας, στο σημείο 5. Προτινόμενος κανονισμός του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή έκτακτης στήριξης εντός της Ένωσης. Πολύ χαίρομαι και για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλο γιατί προεδρεύω εδώ από κοινού με τον συνάδελφο Κλόντο Μωράης που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών που έχουν ε, βέβαια τεράστιο φόρτο εργασίας με διάφορα νομοθετικά ζητήματα. Σήμερα λοιπόν θα μπορέσουμε από κοινού να συζητήσουμε. Επίσης ο Επίτροπος Τηλιανίδης κατάφερε να βρει χρόνο και να έρθει. Παρόλο που τον ενημερώσαμε πριν από πολύ λίγο καιρό. Στις 4 ακριβώς όμως πρέπει να φύγει, γιατί πρέπει να πάει στην Ουκρανία. Όχι, στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Την Τετάρτη πάτε στην Ουκρανία. Εντάξει, Λονδίνο πρώτα. Ναι. Πρέπει και εκεί έχουμε κυκλοφοριακό, ε. πρέπει να φύγει λοιπόν το αργότερο στις 4. Και γιατί λοιπόν του ζητήσαμε να έρθει σήμερα εδώ για να παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη νέα πρόταση κανονισμού για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή έκτακτη στήριξη εντό τη Ένωση. Στι 2 Μαρτίου δημοσιεύτηκε η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια πρόταση στην οποία κατέληξαν μετά από συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Υπουργών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρξει ανθρωπιστική στήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η προσφυγική κρίση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις ήρθαν, συναντήθηκαν με μένα, με συναδέρφους στο φθινόπωρο για να μας πούν ότι παρόλο που υπάρχει χρηματοδότηση για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες στην Τουρκία, στην Ουκρανία, στο Λίβανο κτλ. Δεν προβλέπεται μηχανισμό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προϋπολογισμού για να μπορούν να βοηθηθούν οι πρόσφυγες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρχισαν λοιπόν οι συζητήσεις το φθινόπωρο για αυτό το θέμα και ο Επίτροπος ε, πραγματικά μας άκουσε προσεκτικά και συμφώνησε να δώσει συνέχεια. Τώρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας μία πρόταση για κανονισμό. Η πρόταση αυτή πρέπει να προχωρήσει γρήγορα βέβαια. Βάσει του 122.1 άρθρου της συνθήκης. Δεν είναι ο συνήθις ε, μηχανισμός συναπόφασης αυτός. Θα δώσει λεπτομέρειες ο Επίτροπος πρόκειται για 300 εκατομμύρια το 2016 και 200 το 2017 και 2018. Συμφώνησαν οι χώρες μέλη την Τετάρτη που μας πέρασε και θα επικυρωθεί αύριο από το Συμβούλιο η πρόταση αυτή κανονισμού. Στη συνέχεια θα υπάρξει τροποποίηση του προπολογισμού που θα τεθεί ε, προς έγκριση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε, ε, Επίτροπε, να ξέρετε ότι ανησύχησαν οι συνάδελφοι και ανησυχούν μήπως τα χρήματα αυτά τα βρούμε, τα κόψουμε δηλαδή από αλλού για να τα βάλουμε εκεί, σε αυτό τον κανονισμό. Είναι μια ανησυχία και θέλουμε να μας καθησυχάσετε. Από το τίτλο 3 των πολιτών ε, δημοσιονομικών προοπτικών. Η... Δεν ξέρω, ίσως ε, και ο συμπρόεδρος να έχει κάτι να πει. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ από την Επιτροπή Ανάπτυξης για το γεγονός ότι μας αφιερώσετε το χρόνο για να έχουμε την ανταλλαγή αυτή απόψεων. Σας ευχαριστούμε. Είμαι ευγνώμων δε και προς τον Επίτροπο που με τήρησε ενημερό και σε ό,τι αφορά την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και για το εκτενές έργο σας προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο αυτό όπου η ανθρωπιστική βοήθεια χορηγείται στην καρδιά του προβλήματος. Για μας την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πρόκειται για μια σημαντική συμβολή στην ενοποιημένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προσφύγων και των μεταναστών. Καλωσορίζω λοιπόν ιδιαίτερα στην πρωτοβουλία και θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος, μια και τον Επίτροπο θέλουμε να ακούσουμε. Καλωσορίζω και τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ σας καλώ να θέσετε ερωτήσεις για τον προϋπολογισμό. Να κάνω κάποια ζητήματα να θέσω. Θέλουμε ανταλλαγή απόψεων για έναν κανονισμό του Συμβουλίου, όπως είπε η Λίντα, και συνοδεύεται από έναν διορθωτικό προϋπολογισμό για να υπάρξει μια ξεχωριστή γραμμή σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση για τα ζητήματα τα θαλάσσια για την Ευρώπη από το Ταμείο για τη Μετανάστευση και την ε, αντιμετώπιση των προσφύγων είναι το, τα νέα αυτά πόσα 300 εκατομμύρια το 2016 και 200 εκατομμύρια το 2017 και 2018. Εν ώψη των προτάσεων λοιπόν αυτών, γνωρίζω ότι τα μέλη της Επιτροπής μας θα θέσουν ερωτήσεις στον Επίτροπο για τη χρήση των κοντιλίων αυτών, αλλά και για την νομική βάση, για το πώς θα υπάρξει λογοδοσία. Ξέρω ότι αυτά τα θέματα ετέθησαν στην Επιτροπή μας, αλλά θα ήθελα να διευκρινίσω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για την πρωτοβουλία αυτή και για την συνεργασία με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Κλόντ, λέει η κυρία Αγκέβαν. Και τώρα το λόγο έχει ο Επίτροπος. Thank you so much, of course, for you. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα, και ευχαριστώ για όλα όσα είπες εισαγωγικά. Όντως, από εδώ άρχισαν οι συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ και αγαπητέ κύριε Μωράης. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και σας όλους για την παρουσία σας εδώ προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Όντως χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται παροχή έκτακτης στήριξης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα και αυτή την ανταλλαγή απόψεων, ιδιαίτερα μάλιστα γιατί πρόκειται για μια κοινή συνάντηση με τις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές ανάπτυξης και προστασίας του πολίτη και είναι και η καταλληλότερη στιγμή για να σας παρουσιάσω τα τελευταία νέα όσον αφορά αυτό το νέο μέσο παροχής έκτακτης στήριξης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνεργάτες μου και εγώ, όπως γνωρίζετε, είμαστε σε επαφή με τους πρόεδρους και τους συντονιστές και των δύο αυτών κοινοβουλευτικών επιτροπών όλες αυτές τις τελευταίες μέρες για να σας ενημερώνουμε. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για τα θετικά μηνύματα στήριξης που μας έστειλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την πρωτοβουλία μας αυτή. Και προσωπικά δεν είχα και καμιά αμφιβολία ότι αυτό θα συνέβαινε. Από την έναρξη της εντολής μου, το, από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου δηλαδή, είχα πάντα εξαίρετη συνεργασία μαζί σας και σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Στο τέλος, πριν ολοκληρώσω την ομιλία μου, θα αναφερθώ λίγο και στην Ουκρανία. Διότι θα πάω αυτή τη βδομάδα στην Ουκρανία. Την Τετάρτη το βράδυ θα ταξιδέψω. Λοιπόν, τώρα την ώρα που μιλάμε, πρόσφυγες εξακολουθούν να φεύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες και φτάνουν σε γειτονικέ τους χώρες, αλλά φτάνουν και στην Ευρώπη. Και ο αριθμός τους αυξάνει συνεχώς. Τόσο εκτός Ευρώπης όσο και εντός Ευρώπης. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Θέλω να υπογραμμίσω και πάλι ότι πρόκειται για μια ιστορική υποχρέωση που έχουμε. Πρόκειται για ένα ηθικό καθήκον που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την χωρίς προηγούμενο κρίση. Αντιλαμβάνομαι πλήρως και αναγνωρίζω ότι ζούμε κάτω από έκτακτες συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται και έκτακτες λύσεις, δράσεις. Μήπως θα μπορούσε κανείς πριν από ένα χρόνο να σκεφτεί ότι θα δημιουργούσαμε ένα μέσο παροχής έκτακτης στήριξης εντός της Ένωσης. Όχι. Να όμως που έγινε. Δυστυχώς. Και γιατί έγινε τώρα. Για δύο λόγους κυρίως. Πρώτον, επειδή όλοι βλέπουμε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται όπως περνάνε οι μέρες. Από την αρχή της κρίσης κάποιες χώρες μέλη αγωνίστηκαν να αντιμετωπίσουν αυτή την ανθρωπιστική πρόκληση που είχαν μπροστά τους. Όμως οι ανάγκες μεγάλωναν συνεχώς. Οι προσπάθειες αυτές λοιπόν δεν αρκούν πλέον. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη μάλιστα από τη στιγμή που έχουμε και παράτυπους μετανάστες με το κλείσιμο των ε, διαδρομών προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Πριν από δύο εβδομάδες, ο αριθμός των ε, προσφύγων που ήταν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα ήταν λίγο πολύ 15.000. Σήμερα, ο αριθμός αυτός είναι πάνω από 45.000. Είναι λοιπόν μια μεγάλη πρόκληση να μπορέσουμε να τους προσφέρουμε ε, καταφύγιο, κατάλημα, να ανταποκριθούμε στις βασικές τους ανάγκες. Δεύτερος λόγος. Γιατί έπρεπε να προχωρήσουμε ομαλά, να είμαστε οργανωμένοι, προετοιμασμένοι και ακριβώς αυτό είναι που κάνουμε μέσω του νέου αυτού μέσου στήριξης. Οι ανάγκες των ανθρώπων αυτών μεγαλώνουν μέρα τη μέρα και κάθε μέρα που περνάει είναι μια χαμένη μέρα. Όπως γνωρίζετε, το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας που διαθέτουμε προσανατολίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, μόνο προς τρίτες χώρες. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τον αντίκτυπο της προσφυγικής κρίσης, Έχουμε και τον ε, μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των πολιτών. Έπαιξε κάποιο ρόλο και αυτός ο μηχανισμός, αλλά είναι ένα μέσο που παρόλο που είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι και πανάκια. Γνωρίζετε ότι δημιουργήθηκε ο μηχανισμός αυτός κατά πρώτον και πάνω απ' όλα για να ανταποκριθεί σε περιπτώσεις ε, φυσικών καταστροφών, θεομηνιών, που αντιμετωπίζει η μία ή η άλλη χώρα μέλος. Τώρα όμως έχουμε πάνω από μία χώρα που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, οπότε ο μηχανισμός αυτός έχει φτάσει στα όριά του. Και εξαρτάται πλέον από την εθελοντική συνεισφορά του κάθε κράτους μέλους. Δημιουργήθηκε ο μηχανισμός αυτός για να ανταποκρίνεται σε έκτακτες ανάγκες, όμως δεν φτάνει πλέον, κυρίως κάτω από τις τόσο δύσκολες συνθήκες όπως αυτές που βρισκόμαστε τώρα. Συνεπώς, η ζωή των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και η σωτηρία τους από το θάνατο τον ίδιο είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ένα νέο μέσο, εφόσον δεν μπορούμε με τόσο έχουμε μέχρι τώρα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου καλωσόρισε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει ένα νέο μέσο για να μπορεί να υπάρξει τέτοια παροχή έκτακτης βοήθειας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει λοιπόν της απόφασης αυτής, στις 2 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού. Τώρα λοιπόν θα έχουμε ένα νέο κανονισμό, ο οποίος θα μας επιτρέψει για πρώτη φορά να μπορέσουμε ομαλά να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια και ανακούφιση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέσο αυτό θα μας βοηθήσει να στηρίξουμε και να συμπληρώσουμε τις προσπάθειες των χωρών μελών που αντιμετωπίζουν κυρίως το πρόβλημα. Πρόκειται για οικονομική βοήθεια, για διοικητική βοήθεια, γιατί οι ικανότητες οικονομικές αλλά και διοικητικές των χωρών αυτών έφτασαν στο ωριά τους. Γι' αυτό λοιπόν θα μπορέσουμε μέσω των εταίρων μας την ανθρωπιστική βοήθεια να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη να διαχειριστούν την κρίση. Εννοείται ότι πρέπει να συντονιστούμε με τις χώρες μέλη. Το Συμβούλιο αναμένεται αύριο να υιοθετήσει το νέο αυτό μέσο. 13 μέρες δηλαδή μετά από την πρότασή μας. Η κατάσταση επιτόπου κυρίως στην Ελλάδα, στην Ιδωμένη, αλλά και σε άλλες περιοχές είναι απελπιστική και χειροτερεύει συνεχώς. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε τάχιστα. Η εντολή που δίνουμε αφορά μία τριετή περίοδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει την εφαρμογή της δράσης αυτής μετά το πρώτο έτος. Τώρα, πιο συγκεκριμένα θα αναφερθώ στα ποσά. Η Λίντα ήδη αναφέρθηκε, αλλά θα ήθελα και εγώ να σας εξηγήσω με περισσότερες λεπτομέρειες. Προτείνουμε λοιπόν 700 εκατομμύρια ευρώ να διατεθούν για την επόμενη τριετία. 300 εκατομμύρια θα διατεθούν ήδη για φέτος. Και βέβαια 200 για τον επόμενο χρόνο και 200 για το 2018. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εννοείται ότι συμμετέχουν πλήρως στην ε, λήψη αποφάσεων. Και στηρίζομαι σε εσά προκειμένου να εγκριθεί γρήγορα τροποποιημένος προπολογισμό. Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε την εκταμείευση των πρώτων 100 εκατομμυρίων ευρώ. Και επιτρέψτε μου να είμαι σαφής. Τα χρήματα αυτά είναι επιπλέον από τα χρήματα τα οποία προβλέπονται για τους πρόσφυγες εκτός Ευρώπης. Όταν θα έχουμε στη διάθεσή μας λοιπόν τα κονδύλια, τον προπολογισμό, θα υπογράψουμε συμβάσεις μέσα σε λίγες μέρες με τους εταίρους μας. Τώρα που μιλάμε, οι υπηρεσίε μου συζητούν με τους εταίρους μας, είτε πρόκειται για την υπατή αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, είτε πρόκειται για τη Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση, η Ερθροσταυρό με οργανώσεις, για να δούμε τι προγράμματα μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή βάσει αυτού του νέου κανονισμού θα αρχίσουμε με διάφορες επιχειρήσεις στήριξης, οι οποίες θα αυξηθούν όσο περνά ο καιρός και όσο βέβαια έχουμε και τα απαραίτητα κονδύλια στη διάθεσή μας. Σας διασφαλίζω λοιπόν ότι το μέσο αυτό είναι η προτεραιότητά μας. Θα χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα στις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Θέλω εδώ να τονίσω ότι πρόκειται για έκτακτα μέτρα, για έκτακτους, έκτακτες καταστάσεις και συγχρόνως δεν πρέπει να έχουμε καμία ψευδέστηση. Προκειμένου να υπάρξει πραγματική λύση στο προσφυγικό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες του κακού στις χώρες προέλευσης, στη Συρία, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν και αλλού όπου υπάρχουν σειράξεις. Και γι' αυτό ακριβώς, ως Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια, δεσμεύομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ηγείται της ανθρωπιστικής προσπάθειας που γίνεται για να αντιμετωπιστεί η κρίση στη Συρία και όχι μόνο, και οπουδήποτε αλλού υπάρχουν τέτοιες καταστροφές. Αύριο θα ανακοινώσω συγκεκριμένη χρηματοδότηση για να αντιμετωπιστούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες για την Συριακή κρίση. Και είναι η πρώτη φορά μετά από τη διάσκεψη των δωρητών στο Λονδίνο. Συγχρόνως, θέλουμε να ανταποκριθούμε και σε άλλες ανθρωπιστικές καταστροφές ανά τον κόσμο. Και θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί πολλές φορές υπάρχουν παρεξηγήσεις εδώ τουλάχιστον από αυτά που αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης. Γι' αυτό ήθελα να το τονίσω. Και βεβαίως προσβλέπω στον διαφθορτικό μας διάλογο σε μερικές εβδομάδες προκειμένου να συζητήσουμε την ε, δικιά μας δράση σε όλα τα μέτωπα αυτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της προσφυγικής κρίσης οι χώρες μέλη αντιμετώπισαν οριακές καταστάσεις. Τώρα πρόκειται για την Ελλάδα. Η πίεση στις ελληνικές ακτές είναι πραγματικά δυσανάλογη σε σχέση με τις δυνατότητες που υπάρχουν εξαιτία απλώς και μόνο της γεωγραφικής της θέσης, επειδή βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Εγώ πήγα στην Αθήνα, ήμουν εκεί την ε, Παρασκευή που μας πέρασε και συναντήθηκα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και επανέλαβα την ε, αλληλεγγύη μας απέναντι στην Ελλάδα και συζήτησα μαζί του για να συντονίσουμε την μελλοντική μας δράση. Όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο. Θέλουμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις αυξανόμενες ανάγκες των προσφύγων που φιλοξενούνται στην Ελλάδα και θέλουμε να ανακουφίσουμε τον πόνο τους. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτό είναι το καθήκον μας, η υποχρέωσή μας. Τόνισα λοιπόν στον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη της αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Είπα επίσης στην Ελλάδα και το επαναλαμβάνω και εδώ σήμερα ότι η γενεοδορία των Ελλήνων απέναντι στους πρόσφυγες είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση από όλους μας. Παραδειγματική αυτή η γενοδορία. Μόλις λοιπόν θα έχει εγκριθεί ο προπολογισμό και ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα, σκοπεύω να επιστρέψω στην Ελλάδα. Θα επισκεφθώ εκείνα τα σημεία της χώρας όπου φιλοξενούνται οι πρόσφυγες ή μερικές φορές δυστυχώς πρέπει να πω όπου βρίσκονται εγκλωβισμένοι οι πρόσφυγες κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες όπως την ειδωμένη τώρα. Κάτω από τρομερές συνθήκες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη δικιά της την πλευρά θα διασφαλίσει στήριξη βάσει του κανονισμού και ότι η στήριξη αυτή που θα δοθεί θα συντονιστεί με τις ελληνικές αρχές και με όσους ήδη δραστηριοποιούνται επί τόπου. Και όπως ήδη εξήγησα και στον Έλληνα Πρωθυπουργό και σε άλλους υπουργούς ε, της ελληνικής κυβέρνησης, αυτή η παροχή έκτακτης στήριξης θα δίνεται μέσω των ανθρωπιστικών μας εταίρων επιτόπου. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου τώρα να στραφώ κάπως σύντομα στην Ουκρανία. Θα πάω εκεί την Τετάρτη. Θα είναι η τρίτη μου επίσκεψη στη χώρα αυτή. Το ταξίδι μου στην Ανατολική Ουκρανία, εκεί όπου υπάρχουν οι συγκρούσεις, έρχεται σε κάποια πολύ συγκεκριμένη στιγμή όταν εξακολουθεί να υπάρχει ανθρωπιστικό ζήτημα που όμως δεν αναφέρεται τόσο πολύ πια στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε η κρίση αυτή της Ουκρανίας να γίνει μια ξεχασμένη κρίση. Ένα χρόνο μετά την υπογραφή των συμφωνιών του Μίνσκ, η ειρήνη και η σταθερότητα δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα στα ανατολικά της χώρας αυτής. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να υποφέρουν εξαιτίας της σύγκρουσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει λοιπόν να κάνει έκκληση προς όλες τις πλευρές να τηρήσουν την εκεχηρία. Είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την πολιτική λύση. Και τονίζω και πάλι ότι η Ουκρανία αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική αρρωγή τώρα. Πάω λοιπόν για να επαναλάβω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει απτή αλληλεγγύη απέναντι στους Ουκρανούς. Ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες που πλήττονται περισσότερο και από τις δύο πλευρές της συνοριακής ε, γραμμής. Εκεί ακριβώς είναι που επικεντρώνουμε και εμείς την ανθρωπιστική μας βοήθεια. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται, ενώ μειώνεται η δυνατότητα ανταπόκρισης στην κρίση αυτή δυστυχώς. Θα επαναλάβω επίσης την έκκλησή μας προς όλες τις πλευρές να επιτρέψουν πρόσβαση στους ε, εταίρους που προσφέρουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στο τμήμα εκείνο που δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση. Παρόλο που κάποιες ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν πάρει πρόσφατα την άδεια να συνεχίζουν τα δραστηριότητε τους σε αυτές τις περιοχές, παρόλα αυτά δεν έχουν την ικανότητα να καλύψουν όλες τις ανάγκες επιτόπου. Γι' αυτό λοιπόν επήγει να διευκολύνουμε και την ελεύθερη κυκλοφορία των ίδιων των πολιτών ανάμεσα στην ε, περιοχή την ε, μη ελεγχόμενη από την κυβέρνηση και την υπόλοιπη Ουκρανία. Πάντως η ανθρωπιστική βοήθεια, όπως πάντα, από μόνη της δεν πρόκειται να φτάσει. Χρειάζονται επιπλέον μέτρα για να βοηθήσουμε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους οι οποίοι έχουν μετατοπιστεί, έχουν φύγει από τα σπίτια τους και για να προσφέρουμε κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη για να διατηρήσουν την ελπίδα τους ότι θα έχουν κάποια στιγμή καλύτερες προοπτικές. Οι ουκρανικές πολιτικές δυνάμεις πρέπει να συνεχίσουν επικεντρώνονται στις μεταρρυθμίσεις. Είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη στήριξη από τους Ουκρανούς και από την διεθνή κοινότητα. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβουμε το δικό μας κομμάτι προκειμένου να ανακουφίσουμε τους ανθρώπους που υποφέρουν εκεί. Ακόμα και αν η διεθνή κοινότητα έχει να ανταποκριθεί σε πολλές ανθρωπιστικές έκτακτες ανάγκες, δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στην Ανατολική Ουκρανία. Και πάλι σας ευχαριστώ Λίντα, κύριε Μωράης, για την πρόσκλησή σας και είμαι στη διάθεσή σας τώρα για τα ανταλλαγή απόψεων και για να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε για τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με το νέο μέσο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ας δούμε πόσοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Σημειώνω, Μπίργκιτ, ο κ. Βέντερ, Εν πάση περιπτώσει, ποιος άλλος θέλει για να έχουμε χρόνο. Ο κύριο ε, Βέντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπουμε για το ίδιο το μέσο παροχής ανθρωπικής της βοήθειας ε, στους ε, πρόσφυγες που προσέρχονται στην Ευρώπη. και ε, ως προς τη συνεργασία με τις ε, χώρες ε, διαμετακόμισης. Πώς θα εξεκριβωθεί το νομικό καθεστώς των προσφύγων. Ποιος μηχανισμός δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να διακρίνουμε μεταξύ των διαφόρων ειδών αν θέλετε τύπων ανθρώπων προσέρχονται. Έχουμε οικονομικούς μετανάστες, έχουμε πρόσφυγες Επίσης πώς θα συνεργαστούμε με τις χώρες transit. Ε, αναφερθήκατε και στο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Η Κομισιόν πώς έχει αξιολογήσει τις ανάγκες αυτές. Με ποιον τρόπο τις έχει υπολογίσει. Αναφέρατε κάποια μεγέθη, αλλά πώς τα υπολογίσατε θα ήθελα να ρωτήσω. Μάλιστα, ε, κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να σας πω ότι συμφωνώ απολύτως ότι έχουμε, αντιμετωπίζουμε μια εκτακτή ανάγκη, τη χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα. Όμως γιατί, θα υπογράμμιζα. Και θα έλεγα τα εξής. Εφόσον έχουμε περίπου 3 εκατομμύρια πρόσφυγες στην, στην Τουρκία, διαπραγματευόμαστε όμως ότι μπορεί να πάρει ακόμα περισσότερους. Ταυτόχρονα, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, και λόγω της τάσης διαφόρων κρατών μελών διαβάζουμε το μήνυμα ότι εμείς δεν μπορούμε να αναλάβουμε 3 εκατομμύρια πρόσφυγες, πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό. Αυτό είναι γελίο. Δεύτερον, καθότι υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν αναλαμβάνουν κανενός είδους ευθύνη, δεν δέχονται πρόσφυγες, δεν στηρίζουν οικονομικά, δεν βοηθούν να υποστηρικτεί η κατάσταση στην Ελλάδα και γι' αυτό συζητούμε τώρα για ευρωπαϊκή λύση και εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι απλά αδιανόητο. Με όλους αυτούς τους φράχτες που σηκώνονται παντού, ε, εκατοντάδες χρόνια είχαμε σύνορα στην Ευρώπη, αλλά τέτοιου είδους περίφραξη δεν είχαμε εγκαταστήσει. Επομένως μιλούμε για την ε, απολεσθήσα ε, αλληλεγγύη εντός και εκτός Ευρώπης. Δεν μπορούμε βεβαίως να αφήσουμε στη μοίρα της την Ελλάδα με τους αριθμούς των ανθρώπων που προσέρχονται και οι αριθμοί, επαναλαμβάνω, δεν είναι υψηλή για το σύνολο της Ευρώπης. Αλλά εδώ μιλούμε για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, αλλά αυτά τα χρήματα, αυτή η πόροι δεν είναι καινούργιοι πόροι, είναι πόροι που τους έχουμε μεταφέρει από αλλού. εγώ ε, εξ όσων κατάλαβα από την επανεγκατάσταση προέρχονται οι πόροι και όχι από την ανάπτυξη. Άρα τι σημαίνει αυτό. Ότι εντός του Συμβουλίου εξετάζεται, δεν εξετάζεται πλέον το θέμα της επανεγκατάστασης και η Κομισιόν το ίδιο, την ίδια στάση τηρεί. Επίσης, καθότι σημαντικός αριθμός κρατών, κρατών μελών δεν είναι έτοιμα να δείξουν ελεγγύη. Όλα υποστηρίζονται από τον ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, δηλαδή μακρομπορόθεσμα. πέραν του πρόβλημα, πέραν προβλήματος της Ελλάδος και των προσφύγων, δεν θα υπάρχουν άλλα χρήματα, άλλοι πόροι, διότι δεν επιδεικνύουν αλληλεγγύη τα κράτη-μέλη. Ζητώ συγγνώμη αν μπέρδεψα κάποια μηνύματα με κάποιες ερωτήσεις, αλλά Πραγματικά είναι ανησυχητικά αυτά που βλέπουμε από κάποια κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Η Λόλα Σάντσεθ, Γκουε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο που είναι μαζί μας εδώ σήμερα. Η πρόταση κανονισμού, ε, όπως είπατε, λέτε ότι, όπως είπατε μάλλον, προβλέπει να κατανεμηθεί μέσω οργανισμών και οργανώσεων στο έδαφος και όχι μέσω των κρατών. Αυτό όμως δεν ευθυγραμμίζεται με διάφορες ε, διεθνείς ε, αρχές ε, διαχείρισης, χρηστής διαχείρισης της ανάπτυξης, όπως εκείνες της διακήρυξης του Παρισίου μεταξύ άλλων. Επομένως, η ερώτησή μου είναι τι μέτρα θα αναλάβει η Κομισιόν ώστε να εξασφαλίσει ότι η ενίσχυση αυτή που θα δοθεί θα ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς αρχές αποτελεσματικότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεύτερη ερώτηση πώς θα επιτηρήσετε την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των ε, έργων αυτών. Θα είναι η Κομισιόν θα το κάνει αυτό. Θα γίνει μέσω των κρατών μελών. Ποιος θα προχωρήσει σε αυτήν την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ λέει Πρόεδρος. Έλλη Ευχαριστώ. Λίντα, ε, ευχαριστώ τον κύριο Στυλιανίδη, τον Επίτροπο, προφανώς είναι ένα ε, πολύτιμο μέσο για να αντιμετωπίσουμε την απόλυτη απουσία ε, αλληλεγγύης αυτή τη στιγμή ε, για την ροή μέσω των Βαλκανίων. Πραγματικοί αρκετοί κατήγγυλαν ότι αντιμετωπίζαμε έναν πραγματικό no man's land όπου ένα σωρό οικογένειες είχαν εγκαταληφθεί στην μοίρα τους. Και σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταγγείλαμε μεταξύ άλλων επαλημένως το θέμα και οπότε ε, επιτρέψτε μου να πω καλοδεχούμενο αυτό το έκτακτο μέσο, το μέσο έκτακτης ανάγκης αλλά εν πάση περιπτώσει ας φτάσει η ενίσχυση αυτή στους ανθρώπους που ενεργοποιούνται στο πεδίο δηλαδή τους μη καπαομικρών, δηλαδή εκείνους που εργάζονται άμεσα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς. Τώρα, παρά την εκτακτή ανάγκη και παρά την ε, απόλυτη αναγκαιότητα του μέσου αυτού θα πρέπει η Κομισιόν να μπορέσει να επιτηρήσει την ε, αποτελεσματικότητα της κατανομής των πόρων αυτών και της χρήσεως των πόρων αυτών. Ε, θα ήθελα λοιπόν μια εξασφάλιση ότι θα είμαστε απολύτως ενήμεροι συνεχώς για όλες τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν που θα εφαρμοστούν και θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε, να ελέγξουμε αποτελεσματικά τη ροή των πόρων. Και θα ήθελα μια διευκρίνηση να σας ε, ζητήσω επίσης. Από πού προέρχονται ακριβώς αυτά τα 700 εκατομμύρια που θα διατεθούν. Επίσης, ε, σε σχέση με την Τουρκία, πολύ ανησυχούμε μετά από αυτά που ακούσαμε για τον ε, διάλογο με την Τουρκία, πολλές πτυχές της συζήτησης αυτής μας φάνηκαν απολύτως ε, αντίθετες με την αρχή του νόγο φιλμό, με την αρχή, εν πάση περιπτώσει, των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και συμφωνώ με τους συναδέλφους, με την κυρία Σίπελ. Υπάρχει ένας λόγος που έχουν, έχουμε καθυστερήσει και που αντιμετωπίζουμε την κατάσταση αυτή, ότι τα κράτη-μέλη, αυτό είναι ο λόγο, αρνούνται να αναλάβουν τι ευθύνε του. Και αυτό που αντιμετώπισα και εγώ στη Λαμπεντούζα πριν από ένα μήνα, όλε οι επανεγκαταστάσει αυτέ που υποσχέθηκαν τα κράτη-μέλη και δεν τι υλοποίησαν, αν δεν γίνουν, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Θα πρέπει τα κράτη λοιπόν να αναλάβουν τι ευθύνε και τι υποσχέσει του. Σα ευχαριστώ. Τερέσα Χιμένεθ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο που είναι εδώ μαζί μας. Ζητώ συγγνώμη αλλά ε, αντιμετώπισα κάποια προβλήματα. Να φτάσω από το αεροδρόμιο υπήρχε μια συγκέντρωση. Τέλος πάντων. Ε, στην περασμένη Ολομέλεια του Στρασβούργου ε, μιλήσαμε για την ημέρα της ε, γυναίκας, μιλήσαμε για τους πρόσφυγες γυναίκες, για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αυτές που είναι χωρισμένες από την οικογένειά τους ή από τον άντρα τους και που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερως ευάλωτες μια τραγική, μια δραματική κατάσταση και κατά τη διάρκεια της διαδρομής και κατά την άφηξή τους σε αυτά τα κέντρα, σε αυτά τα τα, στρατόπεδα. Και επομένως η ερώτησή μου είναι αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια για την οποία μιλούμε και γνωρίζω ότι δεν έχουμε πολύτιμες, ε, μάλλον αξιόπιστες στατιστικές αναλύσεις και είναι δύσκολο να δώσουμε ενίσχυση ανάλογα με το φύλλο χωρίς να έχουμε στατιστικές αναλύσεις, αλλά έχετε προβλέψει κάτι για να σκεφτούμε κάποια, ε, κάποια καταλήματα διακριτά ώστε να λάβουμε υπόψη μας αυτές τις ε, γυναίκες με παιδιά που είναι μόνες τους. Και όπως ρώτησαν και οι συνάδελφοι, η κοινή γνώμη, η κοινή γνώμη στη χώρα μας αλλά και αλλού ε, ανησυχεί ιδιαίτερα για την συνάντηση αυτή της 17ης και 18ης ε, αυτά που έχουν διαρρεύσει δεν, ε, δεν ακούγονται πολύ εύσχημα και καλά. Επομένως θα μπορούσατε να μας καθησυχάσετε σχετικά με τη συμφωνία αυτή αν θα βελτιωθεί τι έχει γίνει γιατί μέχρι στιγμής αυτά που έχουμε ακούσει ε, δεν είναι αυτά που ελπίζουμε να ακούμε από την Ευρώπη μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και ο κύριος Μωρές θέλει να θέσει κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα είμαι γρήγορος. Καταρχάς, για τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ εκτιμούμε ιδιαίτερως το ότι πραγματικά χρειαζόμαστε στη χρονική στιγμή αυτή το, το μέσο αυτό. Χαιρόμαστε λοιπόν ε, που το διάθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, η ερώτησή μου είναι η εξής. Το θέμα της νομικής βάσης, το είπα και εισαγωγικά, το έθεσα και στον Αντιπρόεδρο Τίμερμαντς, είναι ε, γενικότερο το θέμα. Το 122 άρθρο, Επίτροπε, βασίζεται στο κεφάλαιο για την οικονομική πολιτική και έχει περιορισμού. Καταρχάς υπάρχει το θέμα του πώς ε, το Κοινοβούλιο μπορεί να συμμετάσχει στι δομέ αυτέ για τη λογοδοσία. Υπάρχει όμω και ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχει κίνδυνο σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό τη ανάγκη, ο οποίο θα μπορούσε ενδεχομένω να διατεθεί σε χώρες σε τέτοια κατάσταση όπως η Ελλάδα. Ήθελα λοιπόν να ελέγξω ποιε είναι οι προθέσει σα, γιατί αυτό αποτελεί θέμα για την Επιτροπή μα και για το έργο μα. Και εν συντομία, γι' αυτό που έθεσε η κυρία Σίπελ, αν το Ταμείο Κατεπίγουσα Ανάγκη ε, ε, προέρχεται από το σχετικό Ταμείο τι θα γίνει, ε, γιατί τι θα γίνει με την μετεγκατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις απαντήσεις σας για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει ταχεία αντίδραση και να υπάρξει συνεχιζόμενη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Και η ΜΚΟ που μας επέστησαν ε, την προσοχή ε, θα πρέπει να συμμετέσχουν και αυτές. Να μην ξεχνάμε επίσης τις άλλες κρίσεις, ε, την Ουκρανία. Αλλά είναι δύσκολο να εξευρεθούν νέα κονδύλια. Αλλά τα κονδύλια θα πρέπει να δαπανηθούν σε αυτούς που τα χρειάζονται πιο πολύ. Και ο λόγος τώρα στην Επιτροπό. Ευχαριστώ, Λίντα. Σας ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις που μου θέσατε. είδα τι εστιαστήκατε σε θέματα προϋπολογισμού ως επιτοπλίστων ασφαλώς. Και εκ παραλίλου εστιαστήκατε στο από πού προέρχονται τα κονδύλια αυτά. Καταρχάς θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής. Η Επιτροπή δεν εγκαταλείπει το σχέδιο κατάσταση. Αντιθέτως, καλούμε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσουν τις αποφάσεις τους σε ό,τι αφορά το σχέδιο κατάσταση. Αναμένω δε και ελπίζω να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα μετά την συμφωνία με την Τουρκία σε ό,τι αφορά το σχέδιο με την κατάσταση. Το θέμα είναι τεχνικής φύσεως, δεν είναι πολιτικό, πιστεύω. Ο σκοπός είναι να χρησιμοποιηθεί ευρωπαϊκός προϋπολογισμός με ευέλικτο τρόπο. για να απαντήσει στις πιο επίγουσες ανάγκες με τα υφιστάμενα κονδύλια. η Επιτροπός Αντιπρόεδρος, ε, κυρία Γεωργίβα, θα απευθυνθεί στην Επιτροπή για τον προϋπολογισμό αυτή την εβδομάδα και θα θέσει λοιπόν την πτυχή του προϋπολογισμού του νέου αυτού μηχανισμού. Θα ήθελα ωστόσο να σας διαβεβαιώσω ότι η πρόθεσή μας ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουμε το σχέδιο με την κατάσταση, σε καμία περίπτωση. Ασφαλώς, τα πρώτα 100 εκατομμύρια δεν θα προέλθουν από την εξωτερική δράση. αλλά από το Ταμείο για τη Μετανάστευση, ΑΦΙΤ, από τα διαστατικά ταμεία ενδεχομένω. Αλλά οι μεταφορές αυτές δεν θα υπονομεύσουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το ταμείο αυτό σε αυτή την κατεπίγουσα κατάσταση. Πρόκειται για μεταφορά για φέτος μόνο. Για το 2017 και 2018 θα υπάρξει μεταφορά από άλλα, από άλλα κονδύλια, όπως για παράδειγμα την ανταπόκριση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή από άλλες πηγές. Να απαντήσω τώρα στα... στη μητρική μου γλώσσα. Για την Τουρκία. Γιατί είναι ευαίσθητο το ζήτημα. Ιδιαίτερα σε τη χώρα μου, την πατρίδα μου, την Κύπρο. Μοιράζομαι μαζί σας πάρα πολλές από τις ανησυχίες σχετικά με τα θέματα της Τουρκίας που έχουν σχέση με την ελευθερία του τύπου και, και ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά την ίδια στιγμή προσωπικά ανήκω σε αυτό που ονομάζεται ρεαλιστική σχολή της πολιτικής. και η εμπειρία μου από το έδαφος και έχω επισκεφθεί την Τουρκία τρεις φορές όπως και τον Λίβανο και την Ιορδανία πολλές φορές μου επιβεβαιώνει ότι για την Ευρώπη η Τουρκία είναι ο key player για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση. και όπως περίπου το κωδικοποιούμε We need them, they need us. Και επειδή είναι αναγκαίο σε αυτές τις συνθήκες να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το κύριο που είναι αυτή η προσφυγική κρίση πιστεύω πολύ σωστά Έχουμε μπει σε αυτό τον διάλογο με την Τουρκία και έχουμε φτάσει στο action plan και στο Turkey facility. Προσωπικά πιστεύω ότι έχεις καλύτερα πολιτικά αποτελέσματα εάν είσαι σε διάλογο με κάποιον παρά να τον απομονώνεις. Δεν θα εμπλακώ στη συζήτηση για το summit αυτή τη εβδομάδα, διότι είναι αποκλειστικό θέμα του Συμβουλίου και δεν έχουμε ακόμη αποτελέσματα για να τα αξιολογήσουμε. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι πολλές οι λεπτομέρειες, μπορούν να γίνουν πολλές συζητήσεις και εκτιμήσεις, αλλά πιστεύω ότι καλύτερα να μιλούμε επί συγκεκριμένου αποτελέσματος παρά να θεωρητικολογούμε. Την ίδια στιγμή όμως, οφείλω ως Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας να πω ότι έχουν γίνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα στην Τουρκία στη βάση του Action Plan και του Turkey Facility. Με τον Επίτροπο Χάν, ο οποίος όπως ξέρετε είναι υπεύθυνο για τον Neighborhood Policy την περασμένη εβδομάδα ανακοινώσαμε projects 100 εκατομμυρίων που έχουν σχέση με το education in emergencies, formal and informal education, and, όπως επίσης και με την διαδικασία cash and voucher, η οποία επεκτείνει μια διαδικασία που ήταν πάρα πολύ πετυχημένη και προσωπικά την είδα στο Καζιάντεπ πόσο ευχαριστημένοι ήταν οι πρόσφυγες εκεί γιατί διατηρούσαν την αξιοπρέπειά τους και την ίδια στιγμή δημιουργούσε καλύτερες συνθήκες και relations between refugees and host communities. Δεν ισχυρίζουμε ότι είναι εύκολο στόχο αυτή η διαπραγμάτευση. Είναι ένα δύσκολο στόχο. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Αλλά οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστές για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αλλιώς η κατάσταση θα, θα χειροτερεύει και θα είναι και εις βάρος αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα εμένα ως Commission for Humanitarian Aid εις βάρος των ανθρώπων που βρίσκονται στη δύσκολη κατάσταση, refugees και migrants, γιατί για μένα ενδιαφέρει αυτός που βρίσκεται στην ανάγκη και πρέπει να τύχει βοήθειας, αλλά την ίδια στιγμή, εάν δεν βρούμε πρακτικά αποτελέσματα, σίγουρα θα έχουμε και προβλήματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουμε προβλήματα στη συνοχή μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναγνωρίσω πολλά από, τα, αυτά που αναφέρατε, ότι περνούμε μια δύσκολη περίοδο. Δεν υπάρχει αφιβολία, υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Όμως, ακόμα και την ιστάτη, πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε ευρωπαϊκή λύση, η οποία να βασίζεται στο European Solidarity. και θέλω να ενισχύσω τις φωνές οι οποίες πιστεύουν ότι δεν υπάρχει λύση με το να χτίζουμε τείχους fences και walls. Δεν υπάρχει τέτοια λύση. Ή θα το λύσουμε όλοι μαζί ή θα αποτύχουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τις πολιτικές διεξόδους και την πολιτική επικοινωνία στον πιο ψηλό βαθμό για να βρούμε το κοινό έδαφος, την κοινή λύση. Έχουμε ακόμα περιθώρια, ευπρόσδεκτη κάθε κριτική, αλλά ας κρατήσουμε και την αισιοδοξία μας, αλλά και την επιμονή μας να βρούμε την κοινή λύση μέσα από, την, από το Common European Solution. θέλω να επαναλάβω ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποτιμήσει το relocation scheme είναι βασικός στόχος πιστεύουμε ότι μετά το επόμενο summit που θα έχουμε συγκεκριμένο αποτέλεσμα θα μπορέσουμε να το επεκτείνουμε. Το ότι μέχρι τώρα δεν έγινε με βάση τις προδιαγραφές που σχεδιάστηκε είναι σωστό και ήταν ένα λάθος, ας το παραδεχτούμε, αλλά ελπίζω ότι μετά το Σάμιτ θα έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε να εφαρμόζεται στην πράξη. Ναι. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποια θέματα που έχουν σχέση με το International Humanitarian Law και σε σχέση με, με τον Geneva Convention. Είχα συνάντηση με τον Φιλίππο Κράντι στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα. Συζητήσαμε όλα τα θέματα, ακόμα και αυτά τα οποία πολύ σωστά ήγηρε ως υπεύθυνο του UNHCR και μοιραστήκαμε την ίδια ευαισθησία απέναντι στους πρόσφυγες και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση αλλά την ίδια στιγμή μοιραστήκαμε και την πεποίθηση ότι υπάρχουν λύσεις μέσα από τα humanitarian principles και το international humanitarian law έτσι ώστε να μπούμε σε μια αποτελεσματική διαδικασία όπου να γίνεται και relocation και resettlement. Σημαίνει θα πρέπει να επιμένουμε στα principles να επιμείνουμε στο humanitarian law, αλλά υπάρχουν λύσει. Να μην νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν λύσει. Αλλιώ, εάν καθυλωθούμε στην άποψη ότι δεν υπάρχουν λύσει, τελικά δεν θα βοηθήσουμε αυτού που έχουν ανάγκη. Και αυτό θα είναι το χειρότερο. Οι πρόσφυγε περιμένουν από εμά λύσει. Δεν περιμένουν συζητήσει νομικού περιεχομένου. Δεν θέλουν να εξαντλούμαστε απλώ σε συζητήσει legalistic approaches or legal issues and matters. Θέλουν πρακτικά αποτελέσματα για τους ίδιους, για τα παιδιά τους, για τις οικογένειές τους. Σχετικά με τα, με τα project στην Ελλάδα και την προετοιμασία που έχουμε κάνει. Όπως είπα οι συζητήσει με την ελληνική κυβέρνηση, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ήταν συζητήσει που διευκρινίσαμε ο καθένα το ρόλο του. Έγινε πλήρη αποδοχή και από τον Πρωθυπουργό και από όλου ότι ναι, υπάρχουν άλλα ευρωπαϊκά φάντς που μπορεί να χρησιμοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση έτσι ώστε ενδεχομένω να δημιουργήσει καταβλισμού προσφυγικού και υπάρχει και χώρο για να μπορέσουν συμπληρωματικά τα humanitarian funds να πάνε μέσω των humanitarian partners έτσι ώστε να είναι συμπληρωματικό προς τις άλλες ενέργειες του ελληνικού κράτους μέσω των διαφορετικών European Funds. Αυτό έχει ξεκαθαριστεί και δεν τίθεται πλέον κανένα ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ερώτηση της αγαπητής φίλης Χιμένες, σχετικά με, τα, με ειδικά project για γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα όντως. Ε, υπάρχουν ανθρωπιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα που they focus on this and we are waiting some project specifically on this very concrete matter Περιμένουμε λοιπόν μια πρόοδο για το θέμα αυτό, φυσικά με συγκεκριμένα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τους ε, ευάλωτους αυτούς ε, ανθρώπους, τις ευάλωτες αυτές γυναίκες και παιδιά. Yes. just, ε, Ναι, και τώρα σε ό,τι αφορά τη νομική βάση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και ιδιαίτερα για τον αγαπητό συνάδελφο, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Λίμπε. το άρθρο 122 επιτρέψει στην Ένωση να δρά σε πνεύμα αλληλεγγύης για να απαντήσει στις κατεπίγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες των προσφύγων στην Ένωση, μέσα στην Ένωση. Και φυσικά να συμβάλλει για να μειώσει, να απαλύνει τον οικονομικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τα εμπλεκομενα κρατημέλη. Η νομική βάση αυτή μας επιτρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα και να εφαρμόσουμε την κατεπίγουσα αυτή αρρωγή μέσω των νομένων οργανώσεων. Γι' αυτό λοιπόν και επιλέξαμε το άρθρο αυτό. At the same time... Εκ παραλίλου, για μας, η βασική ανησυχία είναι η γρήγορη, ταχεία δυνατότητα ανταπόκρισης σε κατεπηγούσες ανάγκες. Αν είχαμε επιλέξει διαφορετική νομιστική βάση, νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση θα υπονομεύαμε αυτό τον βασικότατο στόχο. Γιατί μιλάμε για ένα κατεπήγον ζήτημα και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εκ και ήμουν στο παρελθόν ε, συχνά σε θέση βουλευτή και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνετε σεβαστός και να διαφυλάσσετε ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Τώρα όμως στη χρήση του άρθρου αυτού μπορούμε να πετύχουμε το στοιχείο της κατεπίγουσας δράσης και παράλληλα της διατήρησης των σχέσεων μεταξύ δύο πυλώνων διαθεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, Επίτροπε, λέει Πρόεδρος, για τις ερωτήσεις που απαντήσατε. Αυτά για τα μέλη που, ε, που εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την έλλειψη τέτοιου μηχανισμού. Πέρσι. Και θα σας καλέσουμε και σε άλλες ε, περιστάσεις αργότερα μέσα στο έτο για να απαντήσετε και στα άλλα ζητήματα σε ό,τι αφορά και τι γυναίκε και το καταξύ. Κλόντ, θε να πάρει το λόγο? Ναι, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω και εσά, Λίντα και την Επιτροπή Απασχόληση για την εξαιρετική αυτή συνεδρίαση. Μάλιστα, τώρα λοιπόν διακόπτεται και ολοκληρώνεται η συνεδρίαση, η κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών και θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να μπορέσουν να φύγουν και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Λίμπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μην καθυστερούμε πολύ, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Οπότε, συγγνώμη, όσοι θέλουν να καταλήψουν την αίθουσα, να το κάνουν αυτό γρήγορα, ώστε οι υπόλοιποι να μπορέσουν να καθίσουν. Γιατί έχουμε τώρα ένα σημαντικό θέμα. Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμως μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Πολλοί συζητάμε στην Επιτροπή μας για την ανάπτυξη, εννοείται ότι χρειάζεται μια μακρόπνοη και καινοτόμο στρατηγική για το πόρο και τις επενδύσεις. Είχαμε το γραφό της Επιτροπής, φαντάζομαι το έχετε διαβάσει. Ευχαριστώ για το έργο που έχει γίνει, για την βιωσιμότητα, για τις αλυσίδες εμπορίου, τα διάφορα κριτήρια βιωσιμότητας ε, που έχουν να κάνουν με το εμπόριο. Ο συγητής, ο συντάκτης μάλλον, ο κύριος Χραντήλ, ζήτησε αύριο στις 9 αν είναι δυνατόν να ψηφίσουμε την έκθεσή του. Ελπίζω να συμφωνήσουν οι συνάδελφοι. Στις 9 θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή, Ζαχραντήλ. Εντάξει, ωραία. Αύριο στις 9 ψηφίζουμε λοιπόν αυτή την έκθεση. 64 τροπολογίες είχαμε πολλές τροπολογίες για μια σύντομη, ένα σύντομο κείμενο. Είναι βέβαια σημαντικό το θέμα. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Ζαχραντήλ τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Πρώτον, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους και όλους τους βοηθούς και τους κοιόδης επίσης οι οποίοι συμμετείχαν στην εκπόνηση του κειμένου αυτού. Είχαμε πολλές καρποφόρες συναντήσεις μαζί. Ανταλλάξαμε απόψεις, email και ελπίζω ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια κοινή βάση. Έχουμε 7 συμβαστικές τροπολογίες που ελπίζω να στηρίξουν οι περισσότεροι συνάδελφοι στην Επιτροπή μας. Εντάξει, είναι φυσικό και κατανοητό ότι δεν είναι όλοι απόλυτα ευτυχείς με το κείμενο αυτό. Είχαμε και άλλες τροπολογίες από άλλες ομάδες, αλλά αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι δεν είναι δυνατόν να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Αν μη τι άλλο πιστεύω ότι για τα κύρια θέματα που χειρίζεται η γνωμοδότηση αυτή έχουμε πετύχει κοινοτόπο. Ένα ιδιαίτερο σχόλιο έχω να κάνω όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Και αυτό γιατί ήταν πολύ έντονη η συζήτηση που είχαμε για αυτό το θέμα. Και θέλω εδώ να διευκρινίσω ότι όσον αφορά τη δικιά μου πολιτική ομάδα, που είμαστε υπέρ βέβαια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κατά πόσο πρέπει να είναι υποχρεωτική ή σε θελοντική βάση. Εμείς σαφώς είμαστε υπέρ της εθελοντικής βάσης, γιατί πιστεύουμε ότι οι εταιρείε που επενδύουν στις χώρες μας θα έπρεπε να εγκρίνουν και ήδη το κάνουν, ότι έχουν πρακτικές, έχουν υιοθετήσει πρακτικές πολύ πιο υπεύθυνε. Οι προσπάθειες αυτές όμως πρέπει να παραμείνουν σε θελοντική βάση. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς. Αν όμως εμείς αποφασίζαμε για υποχρεωτικού χαρακτήρα διατάξεις, τότε θα είχαμε περισσότερη γραφειοκρατία, περισσότερο κόστος για τις επιχειρήσεις και κυρίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως γι' αυτό το θέμα που ήταν και το πιο επίμαχο αυτό που συζητήσαμε περισσότερο στις συναντήσεις μας, πετύχαμε έναν καλό συμβιβασμό που είναι η συμβαστική τροπολογία αριθμός 3. Αυτά όσον αφορά τις επεξηγήσεις για αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ και πάλι όλους όσοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα με το κείμενό μας στην αρμόδια επί της ουσίας Κοινοβουλευτική Επιτροπή, την ΙΝΤΑ δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο κύριος Ρούμπικ εκ μέρου του ΕΛΚΑ, μετά ο κύριος Περέιρα. Πολ, εσύ έχεις τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κι εγώ τον συντάκτη, τον κύριο Σαχραντήλ. Όντως, οι συναντήσεις που είχαμε με τους σκιώδη συζήτητες πήγανε πολύ καλά. Οι συμβαστικές τροπολογίες ε, στις οποίες συμφωνήσαμε μας επιτρέπουν την γνωμοδότηση αυτή να την έχουμε ισορροπημένη, κάτι το οποίο θα βοηθήσει και το κείμενο της αρμόδιας επί της επιτροπής. Είναι σημαντικό επίσης οι συνθήκες, οι προϋποθέσεις για τις εμπορικές συναλλαγές να καθορίζονται με σωστό τρόπο οι εμπορικές διευκολύνσεις για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις να επιτρέπουν μια πραγματική εμπορική πολιτική στα πλαίσια του ΠΟΕ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Το διαδίκτυο σήμερα δίνει την ευκαιρία στον κόσμο, στις αναπτυσσόμενες χώρες, να έχει περισσότερες συναλλαγές. Φυσικά και υπάρχουν διαφορές. Αλλά πρέπει να υπάρχει ευημερία για όλους και για τους ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και αυτό θα γίνει μόνο αν υπάρχει μια δικαιοσύνη η οποία λειτουργεί καλά και ένας διοικητικός μηχανισμός που αποφεύγει την διαφθορά και ενθαρρύνει τις επενδύσεις. Εκεί λοιπόν όπου υπάρχουν επενδύσεις, να υπάρχουν προοπτικές για το μέλλον και να μην πρόκειται μόνο για την αύξηση της κατανάλωσης. Η έκθεση αυτή λοιπόν πιστεύω ότι βοηθάει την πρόοδο. Ευχαριστώ λοιπόν και τους και οδησυγητές και όλους όσοι ε, δούλεψαν και βοήθησαν να συνεργαστούμε τόσο καλά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Πέτρος Περέιρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την δουλειά του εισηγητή και την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και η οποία κατέληξε σε αυτές τις ε, συμβαστικές ε, προτάσεις τροπολογίας που έχουμε. Έχουμε μία πρόταση της ε, Επιτροπής Ανάπτυξης που αν εγκριθεί θα είναι μία σημαντική συνεισφορά και αποφασιστική θα έλεγα συνεισφορά. Μιλούμε για την στρατηγική των ε, επενδύσεων αναπτύξεως της Ευρωπαϊκής Ενέσεως για, τους για τα επόμενα έτη και για το πώς η Επιτροπή βλέπει αυτήν τη στρατηγική. Ο δικός μας ρόλος είναι να υπογραμμίζουμε τις πτυχές εκείνες που έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη και να εξασφαλίζουμε την συνέπεια μεταξύ των πολιτικών. στην συγκεκριμένη περίπτωση να εξασφαλίζουμε και τον συντονισμό, αν θέλετε, την ευθυγράμμιση με το θεματολόγιο 2030. Η Κομισιόν έχει διαβιβάσει θετικά μηνύματα, αλλά πρέπει τα έγγραφα στρατηγικής να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη ανάληψη δράσεως. Και για την ε, πολιτική ομάδα υπάρχουν τρία σημεία σημαντικά, τα οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω. Όλα τα μέσα της Αρακής Ένωσης που σχετίζονται με το εμπόριο θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της βιωσίμου ανάπτυξης. Πέραν αυτού, θα πρέπει να προωθούμε ενεργά την συμμετοχική ανάπτυξη. Αυτό θα πρέπει να γίνει επί τη βάση μιας σοβαρής αξιολόγησης, αξιόπιστης αξιολόγησης του αντικτύπου όλων των εμπορικών μέσων, όχι μόνο των μέσων που θεσπίζει με τις αναπτυσσόμενες χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ο αντίκτυπος επί τρίτων χωρών. Και αυτό ισχύει και για τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες. Δεύτερον, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι αυτές οι εμπορικές συμφωνίες, αυτές οι εμπορικές συμβάσεις μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στην ανάπτυξη, όμως αυτό προϋποθέτει ή μάλλον αξίζει να υπογραμμίσουμε τα εξής. Η βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών είναι ουσιαστικό σκέλος πτυχή είναι ένα σημαντικότατο κεφάλαιο, γενικό και οριζόντιο, επί όλων των θεματικών της βιωσίμου ανάπτυξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ε, περιβαλλοντικής προστασίας, της ισότητας των φύλων, για να δώσω μόνο κάποια παραδείγματα. Και τρίτον, θέλαμε να υπογραμμίσουμε το εξής, το οποίο υπάρχει και στις προτάσεις τροπολογίας. δεν γίνεται ρητή μνήα στην Συμφωνία της Κοτονού η οποία θα ολοκληρωθεί το 2020. αξίζει να θυμίζουμε ότι ο διάλογος και η συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ για την μετά την Κοτονού εποχή θα πρέπει συγκεκριμένα να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να έχουμε θετική συνεισφορά στα θέματα της ανάπτυξης ακριβώς για την περίοδο μετά την εκπνοή της συμφωνίας της Κοτονού. Και το λέω αυτό ακριβώς ε, ε, επί της συζητήσεως που έγινε με τις ε, προτάσεις τροπολογίας με τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς λέει η Πρόεδρος, ναι, πράγματι έχουμε διάφορες πτυχές της διαπραγμάτευσης ως προς την Κοτονού. Ο κύριος ο Βάρινεν, θα μιλήσω φιλανδικά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω την αίσθηση ότι ήταν τόσο καλή έκθεση που εγώ δεν υπέβαλα ναι, τροπολογίες. Θα την αποδεχόμουν ως έχει. Ο Λουί Μισελ βεβαίω υπέβαλε κάποιες προτάσεις τροπολογία οι οποίες ελήφθησαν θεωρώ υπόψη επαρκώς στις συμβαστικές. Άνω των 60 έγιναν και συνολικά έχουν βελτιώσει τη σύνταξη του κειμένου. Εκ μέρους τη δική μας ομάδας εγώ μπορώ να σας πω ότι αποδεχόμαστε τις τροπολογίε αυτές. Και στα υπόλοιπα σημεία θα ψηφίσουμε ανεξάρτητα αλλά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για μια πολύ καλή συνεργασία στη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Χόιμπρουκ, ευχαριστώ πάρα πολύ και από δική μου πλευρά. Ε, να ευχαριστήσω για την πολύ καλή ατμόσφαιρα στη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Πραγματικά ήταν πολύ ζωντανέ οι διαπραγματεύσει και θεωρώ ότι η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά πολύ ενθαρρυντική. Ασφαλώ, για εμά του πρασίνου το θέμα είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί φυσικά η εμπορική πολιτική έχει μεγάλε συνέπειε και ιδιαίτερως στι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε του κόσμου αυτού και θα ήθελα να επαναλάβω τις βασικές μας θέσεις. τις οποίες και θα ακολουθήσουμε στην ψηφοφορία. Καταρχάς, η απελευθέρωση εμπορίου είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και στο οποίο ασκούμε κριτική, γιατί θεωρούμε ότι ε, υπονομεύει, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και αυτούς το θέλαμε να τους επισημάνουμε. Δεν είναι αυτόματο δεν είναι αυτόματο ότι με την απελευθέρωση του εμπορίου θα καταπολεμήσουμε τις ανισότητες, τη φτώχεια, την περιθεροποίηση και το καθεξής. Και επισημαίνεται ότι οι χώρες εποφελούνται από την απελευθέρωση μόνο εφόσον ανοίγουν τις αγορές τους πολύ πολύ προσεκτικά και αργά προσαρμοσμένες στις ικανότητες της αγοράς της ίδιας. Άρα η απελευθέρωση δεν σημαίνει αυτόματα κέρδος για τον κόσμο. Στη συνέχεια τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να τοποθετηθούν ε, πιο ψηλά από ότι οι εμπορικές συμφωνίες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να είναι πρώτα-πρώτα αυτά που λαμβάνουμε υπόψη. Και θα πρέπει να υπάρχει πολιτική συνοχή. Και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται δεσμευτικοί κανόνες σε ό,τι αφορά τα εργασιακά πρότυπα, τα περιβαλλοντικά πρότυπα, σε ό,τι αφορά του πραγματικού μηχανισμούς που ισχύουν. Ένα άλλο βασικό θέμα είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η υποχρέωση ε, επεξεργασία των απορριμμάτων για όλη την αλυσίδα παραγωγή και θα πρέπει να σχετή ο παράγοντα αυτό. Και στο σημείο λοιπόν αυτό, στα κρατημέλη μας, χρειαζόμαστε δεσμευτική διάσταση, δεσμευτικό χαρακτήρα σε αυτή την υποχρέωση για τα απορρίμματα και σε ό,τι αφορά τα EPA και θα χρειάζεται πολύ καλύτερη μελέτη αντικτύπου σε ό,τι αφορά τις ε, επενδύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να τα προσμετρήσουμε όλα αυτά. Αυτό συνεπάγεται η πολιτική συνοχή. Δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο τη θεωρία. Θα πρέπει και των εκ των υστέρων να κοιτάμε κάθε φορά πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση, ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες συνέπειες. Και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται σωστή μελέτη αντικτύπου. Αυτά. Εν γέννη, σε ό,τι αφορά τις βασικές μας αρχές, κάναμε και σχετικές τροπολογίες και αυτές, τις, ε, αυτές οι γραμμές θα καθορίσουν και την ψηφοφορία μας αύριο. Ευχαριστώ. Και τώρα από την Γενική Διεύθυνση Trade, από την Επιτροπή, ο κύριος... Από ποια διεύθυνση ρωτάει η πρόεδρος? Δεν, ξέραμε, δεν ξέρουμε. Θα ήταν καλό αν μπορούσατε να διαβιβάσετε στους αδέλφους σας ε, το θέμα αυτό. Ίσως ε, και το θέμα της Συμφωνίας του Κοτονού, αλλά θα επανέλθει το θέμα αυτό μετά την ψήφιση της έκθεσης. Κύριε Σαχραντήλη, θέλει να ξαναπάρει το λόγο, να συνοψίσει. Όχι, σας ευχαριστώ πολύ. Προσβλέπω στην αυριανή ψηφοφορία. Μάλιστα, λοιπόν, ψηφίζουμε στις 9. Πρώτο πρώτο θέμα, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλη τη δουλειά που κάνατε. Προφανώς η συνεργασία ήταν ιδανική και ευχαριστούμε και τους υπαλλήλους που προετοίμασαν του συμβιβασμού. Περνάμε τώρα στο 7. Επιχειρήσεις υπόστηριξη της ειρήνη, δέσμευση που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ΝΑΤΟ και την Αφρικανική Ένωση. Συζητάμε τις τροπολογίε προς την έκθεση, προς την γνωμοδότησή μας μάλλον, ε, για την ε, έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και συγκεκριμένα για την Επιτροπή της ε, ΑΦΕΤ για τα θέματα Άμυνα. Ο κύριος Βάιν είναι εισηγητής μας. Ο κύριος Βαν Όρντεν είναι ο εισηγητής από την ΣΕΝΤΑ. Δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι θα του διαβιβαστούν τα σχόλιά μας. Σε ό,τι αφορά και το άρθρο 54, σε ό,τι αφορά τις ενδεδεμένες επιτροπές. Να δώσω όμως το λόγο στον κύριο Βάινεν Έχετε πολλή δουλειά γιατί και οι επόμενε δύο εκθέσεις, αγαπητοί συνάδελφε, είναι δικέ σα. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα για τι επιχειρήσει υποστήριξη τη ειρήνη. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και ιδιαίτερα μετά τι χθεσινέ επιθέσει και στην ακτή του ελεφάντο του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση του κύριου Φανόρδεν βέβαια ασχολείται κυρίως με τις ειρηνευτικές ε, επιχειρήσεις και το στρατιωτικό σκέλος. Στην δικιά μου γνωμοδότηση πάντως της Επιτροπής μας ασχολούμαι κυρίως με την αναπτυξιακή πολιτική. Το ίδιο και οι συνάδελφοι που συνεργάστηκαν και που έχουν υποβάλει και τροπολογίες αναφέρονται στην αναπτυξιακή πτυχή των επιχειρήσεών μας. Έχουμε τρεις τροπολογίες με τις οποίες φαίνεται ότι συμφωνούν οι πολιτικές ομάδες. Όλοι θέλουμε οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις να αποτελούν μέρος της μεγαλύτερης εικόνας όπου η ανθρωπιστική αρρωγή παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Προσπαθούμε να αποφύγουμε βέβαια τις ένοπλες συγκρούσεις, αλλά η ανθρωπιστική βοήθεια έτσι καλώς έχει να παίξει σημαντικό ρόλο. Υπάρχει και η διαχείριση των κρίσεων για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται σε περιπτώσεις συγκρούσεων. Όταν τελειώνουν οι συγκρούσεις με τη βοήθεια της αναπτυξιακής βοήθειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας μπορούμε να φροντίσουμε να επανέλθει μια ειρήνη διαρκείας και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε στις αναπτυξιακές δράσεις. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες διαφορές στις απόψεις μας, γιατί κάποιοι θέλουν οι ειρηνευτικές ε, επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης δηλαδή, να έχουν κονδύλια όπως εκείνα της αναπτυξιακής βοήθειας. Άλλοι πάλι θέλουν ε, μεγάλη διάκριση ανάμεσα στη μία και την άλλη περίπτωση να χρηματοδοτούνται από διαφορετική γραμμή του προπολογισμού, δηλαδή επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης. Πάντως όλες οι πολιτικές ε, ομάδες συμφωνούν με τις συμβαστικές τροπολογίες και αύριο στην ψηφοφορία είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε πλειοψηφία και να στηρίξουμε τη γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Βέντερ να έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζάχρης δεν είναι εδώ, οπότε εγώ ως συντονιστής έχω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τις επιχειρήσεις υποστήριξης ειρήνης εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία των εισηγητή και για την προσπάθεια που έκανε υπέρ των συμβαστικών τροπολογιών κυρίως τη σχέση ανάμεσα στην ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη και για τον συντονισμό των μέσων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την έκκλησή του στην Αφρικανική Ένωση για δικιά της εμπλοκή. Όντως, είναι πολύ ευαίσθητα αυτά τα θέματα και ότι ο καλύτερος τρόπος να τα αντιμετωπίσουμε είναι στη ρίζα του προβλήματος αλλά συγχρόνως χρειάζεται οικοδόμηση ικανοτήτων και ανθρώπινα δικαιώματα. Οι στρατιωτικοί και άλλες ικανότητες πρέπει να χρησιμοποιούνται υπέρ των ε, πολιτών και ελπίζω η προσέγγιση αυτή να βρίσκεται και στο κείμενο το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Άλλος κανείς για αυτό το θέμα. Όχι. ο κύριος Τάσο Βελάγκα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Δεν έχουμε δει ακόμα εμεί τις συμβαστικέ τροπολογίες, οπότε δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω. Ωραία, ας φροντίσουμε να τις έχουν. Ο κύριος Πινιόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την ΤΕΦΚΟ, έχει να πει κάτι. Ευχαριστώ. Όχι, δεν έχουμε ούτε και εμείς σχόλια. Καλώς. Τίποτα άλλο? Όχι. Ωραία. Θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί και τα σχόλιά μας θα τα προωθήσουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Περνάμε στο επόμενο θέμα του κύριου Βάρινεν, σύσταση σχετικά με την 71η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Αρμόδια είναι η ΑΦΕΤ και είναι και σύσταση προς τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Κύριε Βάρινε, θα σας δώσω το λόγο. Έχουμε 14 τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Με πολύ χαρά ετοίμασα την γνωμοδότησή μου για το θέμα αυτό. Παλιότερα Είχαμε συζητήσει τη δικιά μου έκθεση πρωτοβουλίας όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη. Το σχέδιο αυτό λοιπόν βασίζεται σε μια παλιότερη έκθεση πρωτοβουλίας που είχα κάνει, η οποία βέβαια αναφερόταν περισσότερο σε θέματα αρχής. Τώρα συζητάμε για το μέλλον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Πρόκυψαν κάποια προβληματάκια και πάλι. Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών, για παράδειγμα, μπορεί να γίνει ένα βιώσιμο συμβούλιο. Όταν τα συζήτηγα αυτά στην έκθεσή μου στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης δεν υποστήριζε την ιδέα μου και αυτό με απογοήτευσε για ένα τέτοιο συμβούλιο. Στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων όμως συζητήσαμε και συμφωνήσαμε με έναν τέτοιο στόχο να υπάρξει δηλαδή μια τέτοια αλλαγή στον ΟΗΕ. Να υπάρχει δηλαδή και συμβούλιο για βιώσιμη ανάπτυξη όπως είναι εκείνο ε, το οικονομικό και κοινωνικό. Τώρα, βάσει του μέχρι τώρα έργου, η Ολομέλεια το έχει δεχτεί. Θα έπρεπε να το δεχτεί και εδώ η Επιτροπή μας αλλά κύριοι Πρέντα και κάποιοι άλλοι δεν το δέχονται. Πρότεινα μια συμβαστική τροπολογία της τελευταίας στιγμής, όπου προτείνω να μην αναφέρουμε το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, αν δεν θέλουμε να αλλάξει και να γίνει ένα Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Γι' αυτό και τελευταία στιγμή πρότεινα η πρώτη παράγραφος να συνταχθεί από τον κύριο Πρέντα και αφαίρεσα τη δικιά μου την πρόταση. Θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό γιατί ακριβώς σε αυτήν την Επιτροπή θα έπρεπε να υποστηρίζουμε ένα τέτοιο Συμβούλιο Βιώσιμη Ανάπτυξη πολύ περισσότερο εδώ από ό,τι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία το δέχτηκε όμω. Οπότε ελπίζω αύριο στην ψηφοφορία να το δεχτούμε κι εμείς. Κατά τα άλλα, οι των συναδέρφων ήταν πολύ καλές και όντω βελτιώνουν το δικό μου κείμενο. Πρόεδρος. Έχετε δίκαιο ότι η υλοποίηση της δουλειάς αυτής ε, και το υψηλού επίπεδου πολιτικό αυτό βήμα είναι πολύ σημαντικά για μας. Παρακαλώ, εκ μέρους του κυρίου Πρέντα, ε, Πρόεδρε, ο οποίος θα ήθελε να συγχαρεί καταρχάς τον κύριο Βάρινεν για την σύνταξη του κειμένου και για την ε, συμβαστική τροπολογία της παραγράφου 1. Ο κύριος Πρέντα είναι πολύ ικανοποιημένος που συνεφώνησε ο εισηγητής να υπογραμμίσει περισσότερο την ε, διαδικασία της ε, υλοποίησης και την ενσωμάτωση της ελεύθερης διάστασης της βιωσιμότητας και να συζητηθεί εκ νέου η έννοια του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης. Για το ΕΛΚ είναι πολύ σημαντικό το πλαίσιο του θεματολογίου 2030. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε φιλόδοξες δεσμεύσεις που θα αναλυφθούν προς την υλοποίηση των ESPGs και η ε, ε, θέσπιση συγκεκριμένων δικτών παρακολούθησης. Για την τροπολογία 5 είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει κοινή θέση στην υλοποίηση του θεματολογίου 2030 εν ώψη του υψηλού επίπεδου πολιτικού φόρουμ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ηγηθεί εδώ θα πρέπει να συνδέουμε καλύτερα την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη στα διάφορα σώματα των ΗΕ το οποίο αποτυπώνεται στις τροπολογίες που υπευλήθησαν. Επίσης για την συνοχή της πολιτικής ο κύριος Πρέντα θεωρεί ότι το PCD θα πρέπει να ενισχυθεί με τις δομές των ΗΠΑ. Ε, τέλος, καθότι θα έχουμε συναντήσει υψηλού επίπεδου κατά την Ολομάλια για τις μεγάλες κλίμακες κινήσεις των προσφύγων, ε, θα πρέπει να εστιαστούμε στις ε, οδούς προέλευσης στην ε, κοινωνική ισότητα, στην, ε, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη σταθερότητα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς. Βλέπω κάποιον άλλο συνάδελφο να ζητάει το λόγο. Δεν ξέρω αν ε, η Κομισιόν ή η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θα ήθελε κάτι να πει. Όχι. Μάλιστα. Ο κύριος Βάρινεν έχει την έγκριση της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο μετά τις 9 θα την ψηφίσουμε. Άρα, συνάδελφοι, κινούμαστε γρήγορα. Ήθελα να εξασφαλίσω ότι ο Σκιώδης είναι εδώ για το επόμενο σημείο 9. Την Νέα Συμμαχία για την Ασφάλεια των Τροφίμων και της Διατροφής. Έχει εκδηλωθεί μεγάλο δημόσιο ενδιαφέρον εδώ. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων που έχουμε με την έκθεση και τις ε, τροπολογίες της κυρίας Χόιμπουχ Το Δεκέμβριο είχαμε τις διάφορες ε, θέσεις των ομάδων, το είχαμε συζητήσει και την περασμένη φορά. Έχουμε 15 μονοτροπολογίες. Η κυρία Χόιμπουχ έχει το λόγο, παρακαλώ. Και αν μπορείτε να ειδοποιήσετε παρακαλώ τους ε, σκιώδεις ότι έχουμε προχωρήσει γρήγορα σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίντα. Είπες κάτι που αληθεύει ιδιαίτερος και εμένα αυτή η έκθεση με απασχολεί ιδιαίτερως. Γιατί πρόκειται για το τρόφιμα. Και οι συναδελφοί μου, οι αγρότες ε, όλου του κόσμου, πλήττονται από το θέμα αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν και το προβάλλουμε. Λάβαμε πολλές τροπολογίες. Δεν ήταν πολύ απλό να πετύχουμε συμβιβασμούς και να υπάρξει και μια ισορροπία. Προσπαθήσαμε παρόλα αυτά να καταρτήσουμε ε, πτά συμβαστικές προτάσεις ε, και ευχαριστώ και τους κοιόδους συζητητές. Ε. Να πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, να επενθυμίσω ότι η νέα συμμαχία έχει ως σκοπό τις μεταρρυθμίσεις στην εθνική πολιτική των μεμονωμένων κρατών. Αυτό είναι προβληματικό γιατί από τη στιγμή που περάσει ένα νομοσχέδιο και ψηφιστεί δεν είναι δύσκολο, δεν είναι προφανές και εύκολο να αλλάξει. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω δύο σημαντικούς ε, παράγοντες. Η πρόσβαση στην γη και η πρόθεση του γεωκτήμονα και κατά δεύτερον η βιοπικιλότητα. Καταρχάς λοιπόν σε ό,τι αφορά την ε, πρόσβαση στη γη και την διαφύλαξη της κατοχής της γης. Να υπογραμμίσω το θέμα αυτό, γιατί συχνά υπάρχουν συνθήκες αβεβαιότητας για τους μικρούς παραγωγούς, ιδιαίτερα για τις ε, γυναίκες, των οποίων τα δικαιώματα συχνά δεν αναγνωρίζονται καν και έτσι οδηγούμαστε σε ανισότητες. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, μελέτες ε, που αμφισβητούν τα θέματα σε ό,τι αφορά την πραγματική κατοχή των γεών. Και υπάρχουν διάφορες σχετικές λοιπόν μελέτες που το πιστοποιούν αυτό και από το Πανεπιστήμιο της και από τον ΟΗΕ και μάλιστα στην μελέτη του ΟΗΕ αναφέρεται, αναφέρονται τρεις λόγοι για τους οποίους ε, θα πρέπει να προωθηθούν τα παραδοσιακά δικαιώματα στη χρήση της γης. Καταρχάς, η λογική είναι ότι η πιστοποίηση ε, της ε, ιδιοκτησίας υποτίθεται ότι οδηγεί σε μεγαλύτερη βεβαιότητα. Αλλά αυτό δεν ισχύει απαραίτητα και είναι παραπλαντικό ως παράγοντα, γιατί αυτό ουσιαστικά έχει να κάνει με την πώληση. Ουσιαστικά η γη γίνεται εμπορικό αγαθό. Και αυτό οδηγεί λοιπόν ουσιαστικά σε μεγαλύτερε αβεβαιότητε σε ό,τι αφορά την δεκτησία Η επιστοποίηση αυτή ε, είναι πιο ακριβή, οι πιο πλούσιοι έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στη διαδικασία αυτή και για όσους δεν έχουν τέτοιες, ε, δεν έχουν στην κατοχή τους ε, γη, ουσιαστικά η διαδικασία αυτή είναι και πολύ ακριβή και δυσκίνητη και δυσνόητη. Σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να αγοράσουν, όταν παίρνουν δάνεια δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν. Και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη ανασφάλεια Άρα, σε ό,τι αφορά το land titling, θα θέλαμε να το ε, βάλουμε με ένα ερωτηματικό. Τα θέματα λοιπόν πιστοποίησης ε, της κατοχής γης ε, ουσιαστικά οδηγούν σε όξυνση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών και αυτό το πιστοποιεί και μια σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή και επίσης οδηγεί σε κερδοσκοπία των αλλαδαπών επενδυτών και αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε κάποιες περιπτώσεις σε μεγαλύτερη συγκέντρωση των γεών. Στις χώρες δε που υπάρχει ήδη ανισότητα στην κατοχή της γης, οι διαφορές αυτές οξύνονται. Και δεν μιλάμε μόνο για την πιστοποίηση της κατοχής, αλλά και για το δικαίωμα χρήσης της γης και πρόσβαση σε τέτοια, σε τέτοια σε, στη γεωκτησία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα δικαιώματα αυτά χρήσης, Είναι σημαντικό αυτό και για τους ε, εκτροφείς και για τους αλληλείς. Το συμπέρασμα λοιπόν για μένα, για το τμήμα αυτό της έκθεσης, είναι ότι η πιστοποίηση αυτή της γεωκτησίας πρέπει να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπονομεύονται τα δικαιώματα των μικρών καλλιεργητών προκειμένου να δημορφώσουν ε, μια αξιοπρεπή εκμετάλλευση. Άρα χρειάζονται αυστηροί κανόνες, αυστηρή, αυστηρά πρότυπα για τη μεταφορά της γης και σε ό,τι αφορά τους επενδυτές, προκειμένου τελικά να μην υπάρχει μεγαλύτερη φτώχεια. Και τα δικαιώματα ευημερίας θα πρέπει σίγουρα να υπογραμμιστούν. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη γη η νέα συμμαχία θα πρέπει να διεξαγάγει Μάλλον θα πρέπει να περάσει από μελέτη αντικτύπου σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα πρόσβαση στη γη. Θα πρέπει να βλέπουμε πάντα ποια είναι τα, ποιες είναι οι συνέπειες της κάθε απόφασης και αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θα πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένος και να συνενεί. Και αυτό αναφέρεται και στις εθραντικές ε, κατευθυντήριες γραμμές ε, τις οποίες έχει δεσμευθεί αυτή η νέα συμμαχία ότι θα εφαρμόσει. Είναι σημαντικά λοιπόν αυτά τα στοιχεία που αναφέρονται στην έκθεση γιατί συνάπτουν και με τις διεθνείς υποχρεώσεις. Δεν επικαλούμαστε μόνο το πράσινο όραμα, όχι. Επικαλούμαστε και αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στις διεθνείς συμβάσεις. Τώρα, για τους σπόρους θα πρέπει να μετρηθεί τα δικαιώματα του καλλιεργητή προκειμένου να μπορούν ελεύθερα να πολλούν και να χρησιμοποιούν τους σπόρους. 90% των αγροτών στην Αφρική εξαρτώνται από την ελεύθερη χρήση αυτών των σπόρων και χρειάζεται λοιπόν ε, ο τοπικός, η τοπικός πλούτος ε, σπόρων και η ε, προσαρμοσμένοι και αυτό σε τιμές τους οποίους ε, τις οποίες δεν μπορούν να πληρώνουν οι αγρότες. Αυτό φυσικά εξυπηρετεί και την βιοποικιλότητα και αποτελεί και μια βάση για την ε, επισητιστική αυτάρκεια. Η Νέα Συμμαχία μιλάει και για την ε, οδηγία του 91 σε ό,τι αφορά τις ανεπίσημες πρακτικές εμπορίας σπόρων τις οποίες και σκοπεύει να τις ε, καταργήσει. Αλλά η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι σπόροι προσαρμοσμένοι σε τοπικό επίπεδο. Η έκθεση αυτή δεν θα πρέπει να θέσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε ό,τι αφορά και το σκοπό της βιοπικιλότητας. Ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω τα δύο αυτά σημεία, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί αφορούν ασφαλώ την επιστημική ασφάλεια, όχι μόνο την ε, εξασφάλιση επαρκών θερμίδων, αλλά και την εξασφάλιση μίας ε, υγιούς και διαφοροποιημένης διατροφής. Και αυτό το εξασφαλίζουμε και με την ε, σωστή καλλιέργεια. Προς την κατεύθυνση αυτή σημαντικά είναι δύο στοιχεία, η γη και οι σπόροι. Θεωρώ ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον το έργο και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν και μας βοήθησαν. Να ευχαριστήσω δε και για την καλή ατμόσφαιρα κατά την διαπραγμάτευση, ακόμα και αν δεν είναι εδώ οι συνάδελφοι. Thank you, Maria. Ευχαριστούμε, Μαρία, για όλη αυτή τη δουλειά. Ποιος θα ήθελε να έχει το λόγο. Ο κύριος ε, Βάρινεν. Πρόεδρε. Δεν είμαι σκιώδης ε, εισηγητής εδώ, αλλά έχω υποβάλει κάποιες ε, προτάσεις τροπολογίας, θα ήθελα να τις ε, συζητήσουμε. Το σχέδιο είναι πολύ καλό. Και οι συμβαστικές που συζητήθηκαν φαίνονται επίσης να είναι πολύ καλές. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι τρεις δικές μου στο 104, 105 και 106 Τις βρίσκω όμως σημαντικές και θα ήθελα να σας εξηγήσω γιατί. Ε, θεωρώ ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος. Όταν έχουμε μεγάλες κλίμακες επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες, σημαντικά δηλαδή έργα, τα οποία θα οδηγήσουν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ίσως προβλήματα, θα πρέπει να ταρίσουμε τέτοια στάση ώστε να υποστηρίζουμε τις ε, υφιστάμενες μικρής κλίμακος εκμεταλλεύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να κινηθούμε μέσω εθνικών γεωργικών και αγροτικών ταμείων που δίνουν, παρέχουν ενισχύσεις ε, στους ε, αγρότες, τουλάχιστον στις σκανδιναβικές χώρες ήταν ένας τρόπος υπό τον οποίο πετύχαμε βιώσιμη γεωργία και έχουμε εμπειρία με αυτό. Θα πρέπει επίσης να προσέξουμε την ε, εκπαίδευση και κατάρτιση των μικρών αυτών ιδιοκτητών και καλλιεργητών ώστε να επιτύχουν ένα υψηλότερο βιωτικό επίπεδο και υψηλότερη παραγωγικότητα. Και τέλος, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε τις επαγγελματικές και οικονομικές ενώσεις των καλλιεργητών, των γεωργών, την συνεργασία που έχουν συστήσει, όπως και τους συνεταιρισμούς, ώστε να λαμβάνουν και σπόρους και εξοπλισμό σε ανταγωνιστικές τιμές και ώστε να υποστηρίζονται και ως προς το μάρκετινγκ των προϊόντων τους. Και σε αυτό το τομέα είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα και στο μάρκετινγκ και στη μεταποίηση. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα υποστηρίξουμε τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, για παράδειγμα, ή στην Αφρική και να ανησυχούμε για τόσο μεγάλης κλίμακος ε, παραγωγή που θα είχε σημαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτω... δεινές επιπτώσεις. Ελπίζω λοιπόν να ληφθούν υπόψη οι τρεις μου αυτές ε, προτάσεις και οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων επίσης ενδεχομένως να τις υποστηρίξουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ε, Νόιζα. Ευχαριστώ. Ε, η εκπροσωπώ των, Δίκα ο οποίος ε, ζητάει συγγνώμη για την απουσία του. Ο σκιώδης μας θα ήθελε να συγχαρεί την Μαρία για την δουλειά αυτή και τον συντονισμό και την συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών ομάδων που επέτυχε. Νομίζω ότι έχουμε συμβιβαστικές που υπογραμμίζουν ότι καταρχάς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπογραμμίσει τα όποια, να καλύψει μάλλον τα όποια κενά και στη διαφάνεια και στη διακυβέρνηση ώστε αυτά να γίνουν συμβατά με τους ε, στόχους της βιωσίμου ανάπτυξης θα πρέπει επίσης να προαγάγουμε βιώσιμη χρήση της γης, πρόσβαση των μικροϊδιοκτητών και των μικροκαλλιεργητών και για την ιδιοκτησία του γενετικού υλικού. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την τοπική και περιφερειακή αγορά ώστε να έχουμε δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας και εργασιακών δικαιωμάτων θα πρέπει να έχουμε επίσης αυξημένο έλεγχο επί των ε, εταιρικών συνεργασιών δημοσίου ιδιωτικού δικαίου ώστε να είναι ένα διαφανές εργαλείο ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το 100% του δυναμικού μας και υπό την έννοια αυτή ε, θα θέλαμε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των γυναικών της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών αρχών και των τοπικών κοινοβουλίων στην υλοποίηση των αρχών της συμφωνίας πλαίσιο. Είναι σαφές ότι το μέλλον της Αφρικής είναι στα δικά τους χέρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τους βοηθήσει και να τους ενισχύσει προς την ασφάλεια των τροφίμων και την βιώσιμη ανάπτυξη. Εκ μέρους του Ενρίκε θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές για την συμμετοχή τους και τη συνεργασία τους. Ο Ενρίκε είναι βέβαιος ότι θα έχουμε μια ισχυρή κοινή θέση μετά την ψηφοφορία αύριο. Ευχαριστώ και πάλι Μαρία. Θέλει κανείς άλλος το λόγο για αυτό το θέμα. Κύριο κύριος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, εσείς. Σας είδα όταν μπαίνατε, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, περιμένουμε να είσαστε σε θέση, να πω μόλις μπήκατε. Εντάξει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, Θέλουμε να συγχαρούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ανέλαβε την πρωτοβουλία για την έκθεση αυτή όσον αφορά την επισυταστική ασφάλεια και τη νέα συμμαχία για τη διατροφή. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε και από τις Ηνωμένε Πολιτείες σε κάποιο έτσι προεδρικό στυλ. Πάντως το έργο του Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και για να εντοπιστούν τα δυνατά σημεία της νέας αυτής συμμαχίας, αλλά και οι αδυναμίες της, πάνω στις οποίες πρέπει να δουλέψουμε. Δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιγράψουμε στην Αφρική τα ίδια μοντέλα, τα αναπτυξιακά που έχουν εφαρμοστεί σε άλλα μέρη του κόσμου. Αυτό είναι κάτι που το λέμε και εμείς στην Επιτροπή ξανά και ξανά. Το άλλο είναι ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες ρήτρες ασφάλειες κάθε φορά που προωθούμε επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα προς ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα προς αφρικανικές χώρες. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ σημαντικό το θέμα της πρόσβασης σε γη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με τις υπεύθυνες επενδύσεις στην Γεωργία. Ο λόγος που θέλουμε αυτές τις δύο ρήτρε ασφάλειας είναι γιατί οι επενδύσεις στη Γεωργία πρέπει να προστατεύουν εκτός από την κοινωνική διάσταση και την περιβαλλοντική. Και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, είναι η λογοδοσία. Κάθε φορά που μιλάμε για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων. Εσείς ζητάτε περισσότερη λογοδοσία. Εισακουστήκατε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι συζητούμε και εμείς και συζητιέται και σε αυτό το κτίριο είναι μια άλλη πρωτοβουλία για χρηματοδότηση της γεωργίας. Στόχος είναι περισσότεροι πόροι, περισσότερα κονδύλια για τη γεωργία. Έχουμε τρεις επιλόνες εδώ. Ο πρώτος είναι η αναγνώριση της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων των αγροτών κάθε φορά που μιλάμε για ιδιωτικές επενδύσεις. Πρέπει να είναι ο πρώτος επενδυτής και να μπορούν να παίξουν ρόλο και να συζητήσουν. Ο δεύτερος πυλώνας είναι να μπορεί να επενδύει ο ιδιωτικός τομέας και το τρίτο που έχει να κάνει με τη λογοδοσία είναι μια πρωτοβουλία που έχουμε αρχίσει που έχει να κάνει με την αξιολόγηση. Δηλαδή οι δωρητές όταν στηρίζουν ιδιωτικές επενδύσεις πρέπει να γνωρίζουν πριν γίνει η επένδυση ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της επένδυσης στην ε, αλυσίδα αυτή τη διατροφική με μάλιστα ποσοτική έκφραση. Να ξέρουμε δηλαδή πόσοι αγρότες θα συμμετέχουν, τι σημαίνει αυτό για αυτούς. Ή θα έχει επιπτώσεις η επένδυση αυτή στον τρόπο εργασίας. Χρειάζεται κάποια αλλαγή. Και μπορώ εδώ να σας πω ότι για αυτή την πτυχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ηγετικό ρόλο μεταξύ όλων των φορέων. Αναγνωρίζω πλήρως την προσθέμενη αξία των συστάσεων της έκθεσης αυτής και θα τις λάβουμε υπόψη μας τις συστάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Να υπενθυμίσουμε στους συναδέρφους, γιατί τον Απρίλιο μόνο θα ψηφίσουμε, ότι έχουμε μία μελέτη για την ε, αυτή συμμαχία. Το τμήμα έρευνάς μας ε, την έχει την ε, έρευνα αυτή ακόμα, οπότε αν θέλετε να ενημερωθείτε, κοιτάξτε. Ωραία. Θέλει κανείς να προσθέσει κάτι, συγκήτρια. Ναι, καταρχάς θα ήθελα να επαναλάβω ότι συμφωνούμε πάρα πολύ, συνάδελφε, με τις ε, τροπολογίες σας, τις οποίες θα ψηφίσουμε ασφαλώς όλες και θα τις υποστηρίξουμε. Επισημάνονται πολύ σημαντικά στοιχεία. Χαίρομαι δε με τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως με το γεγονός ότι δεν θέλετε να επαναλάβετε την πράσινη επανάσταση της Ασίας στις δεκαετίες του 60 Είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι έχουμε διδαχθεί από το παρελθόν. Χαίρομαι που αναφερθήκατε και στα ενθαρρυντικά πρότυπα του ΟΗΕ για την πρόσβαση στη γη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό και περιλαμβάνονται σχετικές αναφορές και στην έκθεση για τις υπεύθυνε τώρα ε, επενδύσεις και στο κοινωνικό και στον περιβαλλοντικό τομέα. Και εδώ νομίζω ότι είμαστε σύμφωνοι. Εγώ θα ήθελα να είναι βέβαια δεσμευτικά αυτά, όχι α, προαιρετικά. Και θα πρέπει να ορίσουμε το τι επιθυμούμε στον τομέα αυτό. Το ίδιο ισχύει και για την υποχρέωση α, λογοδοσίας, ό,τι ισχύει και για τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να ισχύει. Αν δεν υπάρχουν δεσμευτικές ε, δεσμευτικά πρότυπα ουσιαστικά δεν θα εφαρμοστούν ιδιαίτερα και αυτό δεν μπορεί να αποτελεί στόχο μας. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους και αν υπομονώ να δω τι θα γίνει και τον Απρίλιο που θα έχουμε την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Πολλές ε, οι τροπολογίες, άρα πολύ και η δουλειά για την ε, κατάρτιση συμβαστικών προτάσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 20 Απριλίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πήρε το λόγο γιατί πάμε πολύ γρήγορα και προχωράνε γρήγορα τα θέματα σήμερα το απόγευμα. Και αυτό επειδή ο Επίτροπος αναγκαστικά έπρεπε να φύγει στις 4. Στο 16 για την ε, εκλογή των ε, αντιπροσώπων στην ε, για την αποστολή στην Ουγγάντα σε ό,τι αφορά τις... ε, την Επιτροπή Παρατήρησης Εκλογών. Νομίζω ότι περιμένουμε και τον ε, αρμόδιο. Την πρέσβη. της Ουγγάντα. Δεν ξέρω πότε θα καταφτάσει, λέει η Πρόεδρος. Ωραία. Θα αρχίσουμε σε λίγα λεπτά. Είναι στο κτίριο από ό,τι φαίνεται. Ο κύριος Λάινεν θα είναι εδώ όπου να είναι. Σε λίγα λεπτά θα αρχίσουμε πάλι.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 είμαστε λίγο νωρίτερα από το προβλεπόμενο, οπότε συνάδελφοι θα έρθουν σιγά σιγά. Είμαστε στο σημείο 10, αποστολή παρατήρησης εκλογών στην Ουγγάντα. Στα μέσα Φεβρουαρίου, πριν από ένα μήνα, λοιπόν, ήταν η αποστολή αυτή. Έχουμε τον κύριο Κούκαν, ο οποίο ήταν επικεφαλή των παρατηρητών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και τον Γιώ Λάινεν, ο οποίο ήταν πρόεδρο αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συνάδελφοι μπορεί να γνωρίζουν ότι ο πρόεδρο Μουσεβένη επανεκλέγει για την ε, πέμπτη φορά το 86 ήταν η πρώτη φορά που ανέλαβε τα προεδρικά καθήκοντα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κούκαν, θα μας εξηγήσετε το πλαίσιο, θα μας πείτε τι έγινε εκεί. Ξέρω ότι υπάρχουν ανησυχίες, η Επιτροπή μας το ξέρει δηλαδή όσον αφορά την Ουγκάντα. Υπάρχουν ζητήματα εκεί, πώς εσείς βλέπετε ότι έγιναν οι εκλογές, αλλά και γενικότερα θέλουμε την άποψή σας και για την αναπτυξιακή κατάσταση της χώρας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και για την πρόσκλησή σας. Θα αρχίσω ευχαριστώντας την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για την τόσο καλή συνεργασία που είχαμε και για την προετοιμασία της αποστολής αυτής παρατηρητών. Ευχαριστώ επίσης και τον πρέσβη Σμιτ που ήταν επικεφαλής και τον κύριο Γιολάινεν που ήταν πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλα αυτά δεν τα λέω έτσι για να πω ωραία λόγια, να είμαι καλός διπλωμάτης. Όχι. Πράγματι, πολλά γεγονότα καταδεικνύουν ότι τα λόγια αυτά ταξίζουν τις ευχαριστίες αυτές. Τώρα, για την ίδια την αποστολή. Ήταν η τρίτη στην Ουγκάντα μετά από το 2006 και το 2011 που είχαμε άλλες δύο. Και δείχνει το γεγονός αυτό την ε, υποχρέωση που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ενίσχυση της δημοκρατίας εκεί. 28 Σεπτεμβρίου που μας πέρασε λοιπόν, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, παρακολουθήσαμε όλη την εκλογική διαδικασία όπου συμμετείχαν 130 παρατηρητές. Αυτό ήταν το πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες διεθνείς αποστολές παρατήρησης της Commonwealth, κοινοπολιτείας δηλαδή, της Αφρικανικής Ένωσης, που πάνε εκεί λίγες μέρες πριν. Εμείς ήμασταν εκεί καθόλου τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και είναι ακόμα εκεί συνάδελφοι. Και θα σας πω γιατί. Εξακολουθούμε να έχουμε τον ε, νομικό μας αναλυτή, τον εμπειρογνώμονα, τον τα την εμπειρογνώμανα μάλλον την Ιταλίδα, η οποία συμμετέχει σε μία διαδικασία ε, που ζήτησε η κυρία Μπαβάζη από την αντιπολίτευση. Τώρα, πολιτικά μιλώντας στην Ουγκάντα, ήταν οι τρίτες πολυκομματικές εκλογές. Και βέβαια υπήρξαν πολλές ε, διαφορές ανάμεσα στα κόμματα και το κράτος. Ο κύριος Μοζεφένη από το κίνημα Εθνικής Αντίστασης βρίσκεται στην εξουσία για 30 χρόνια. Ήταν η πέμπτη, για την πέμπτη θητεία του ήταν υποψήφιος. Υπήρχαν 8 υποψήφοι για τις προεδρικές αυτές εκλογές, τρεις πιο γνωστοί, ο Μουσέβενη, ο κύριος Κίτσα Πεζίγκε από το Φόρουμ της Δημοκρατικής Αλλαγής και η Αμάμα Μπαμπάζη, που... ο Αμάμα Μπαζάντη, που ήταν εταίος πρωθυπουργός και πήρε πολύ χαμηλά αποτελέσματα σε σχέση με αυτά που περίμενε. Οι αρχικές ανησυχίες σχετικά με τις εκλογές αυτές είχαν ε, να κάνουν με παραβιάσεις στην εκλογική διαδικασία, με το να μην μπορούν να έχουν ίση πρόσβαση στα μέσα ενημέρωση όλοι οι υποψήφοι και για το κατά πόσο θα ήταν ε, έγκυρο το μητρό των ε, ανθρώπων που μπορούσαν να εκλέξουν. Την ημέρα των εκλογών τώρα συμμετείχαν οι υποψήφοι και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και οι άνθρωποι που πήγαν να ψηφίσουν έκαναν τεράστιες ουρές στα εκλογικά κέντρα την ημέρα των εκλογών. Για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία της Ουγκάντα έγινε και συζήτηση με όλους τους υποψηφίους και τον Μουσεβένη και τους άλλους. Σε εμά στις δικές μας χώρες θεωρείται κάτι φυσιολογικό, αλλά εκεί είναι κάτι που εκτιμούν όλους ιδιαίτερος. Από την άλλη πλευρά, πλευρά βέβαια, το κίνημα εθνικής αντίστασης οδηγήθηκε σε μια άδικη εκστρατεία. Δημιουργήθηκε μια, ένα κλίμα εκφοβισμού τόσο για τους υποψήφιους της αντιπολίτευσης όσο και για τους εκλογείς. Ούτε ε, τα χρήματα τα οποία δικαιούταν δεν μπόρεσαν να πάρει όλα. Τώρα για την ε, ανεξαρτησία της εκλογικής επιτροπής. Άργησε να φέρει το εκλογικό υλικό την ημέρα των εκλογών σε διάφορες περιφέρειες. Κυρίως στην Καβάλα, την πρωτεύουσα. Και έτσι μειώθηκε η δυνατότητα για πολλούς εκλογείς να καταγράψουν την ψήφο τους. Επίσης εμποδίστηκε και η πρόσβαση στα μέσα ενημέρωση, στα κοινωνικά μέσα, άρα υπήρξε πρόβλημα με την ελευθερία έκφρασης. Ο πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής ανακοίνωνε τα προκαταρτικά αποτελέσματα. Τα πολιτικά κόμματα εξακολουθούσαν να μαζεύουν στοιχεία από τους δικούς τους. Τότε η ε, αστυνομία τα βάλε με το FDC, το κόμμα του Μπετζίκε και τον ε, ίδιο τον πρόεδρο. Υπήρξε λοιπόν παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης. Η εκλογική επιτροπή είναι ανεξάρτητη. Αλλά την εντολή της την ερμηνεύει παρακολουθώντας τα τεχνικά στοιχεία. Δεν υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις αποφάσεις της και δεν ενημερώνει τους εκλογείς και όσους προσφεύγουν όσον αφορά διάφορα στοιχεία κλειδί στην διαδικασία και δεν το κάνει αυτό σίγουρα με κατανοητό τρόπο. Σωστό επίσης θα ήταν να παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα με κατανοητό τρόπο. Άρα λοιπόν οι παρατηρητές μετά τις εκλογές υπέβαλαν μία δήλωση με την οποία θα την εκλογική επιτροπή να δημοσιεύσει χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα από κάθε εκλογικό τμήμα όσον αφορά τις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές online και να υπάρχουν και σκαναρισμένα τα αποτελέσματα. Ο πρόεδρος Μουσεβένη ανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών αυτών Ο Μπαμπάση βρέθηκε πολύ πίσω με 1,39%. Η κατάσταση στη χώρα τώρα μετά τις εκλογές ποια είναι. Μα απασχολεί το θέμα του κύριου Βεζίγκη, ο οποίο αυθαίρετα κρατεί τα κόμμα, χωρίς να του έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία. Υπήρξε εκφοβισμό των συναδέλφων του στο κόμμα, κάτι το οποίο μπορέσαμε με σαφήνεια να καταγράψουμε. Οι υπηρεσίες ασφάλειας επίσης όλο και περισσότερο είναι παρούσες για να εμποδιστεί κάθε διαμαρτυρία. Τα επόμενα βήματα. Ο κύριος Μπαμπάζη και οι δικοί του υπέβαλαν προσφυγή στον το δικαστήριο για να αμφισβητήσουν την δικαιότητα των αποτελεσμάτων των εκλογών αυτών. Κατά του εκλεγμένου Προέδρου, του Μουσεβένη και κατά του Γενικού Εισαγγελέα και της Εκλογικής Επιτροπής με 28 παραβάσεις και παράνομες πρακτικές κατά την εκλογική προεκλογική περίοδο από τον πρόεδρο Μουσεβένη και την εκλογική επιτροπή, μεταξύ άλλων δωροδοκίες, ψεύτικες δηλώσεις σε βάρος άλλων υποψηφίων, ανάμειξη στις εκλογικές δραστηριότητες, χρήση κυβερνητικών πόρων χωρίς να επιτρέπεται και τέλος καθυστέρηση του εκλογικού υλικού στα εκλογικά κέντρα. Περιμένουμε την απόφαση των νότο του δικαστηρίου βέβαια που θα αποφασίσει στις 31, ε, στις 31 Μαρτίου. Στις 18 Απριλίου θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα. Τώρα να μην αναφερθώ στις οικονομικές δυνατότητες, στο μέλλον ε, της χώρας. Είναι μια πολύ σημαντική αφρικανική χώρα η Ουγγάντα αναπτύσσεται με διάφορα προβλήματα εξαιτία της θέσης της χώρας. Έχει πάρα πολλούς νέους η Ουγγάντα. Οπότε η εκπαίδευση, η απασχόληση είναι σημαντικά ζητήματα. Οι οικονομικές δυνατότητες υπάρχουν τεράστιες για την ανάπτυξη της χώρας. Όμως η κυβέρνηση πρέπει να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα και να θέσει προτεραιότητες για το μέλλον της Ουγκάντα. Ευχαριστώ. Okay, thank Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κούκαν και θα ήθελα να πω συγγνώμη προς ε, τον πρέσβη που αρχίσαμε πριν καταφτάσατε. Ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα με τις διαδηλώσεις των αγροτών. Καλώς ορίσατε λοιπόν ε, κύριε πρέσβευτα και καλώς ορίζουμε και τον γραμματέα σας να ακούσουμε και τον Γιώργο Λάιναν, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ε, Αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Η Αποστολή παρατηρήσεις των Εκλογών της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πολύ καλατεχούμενη στην Ουγγάντα λίγες μέρες πριν και την ίδια την ημέρα της εξαγωγής των εκλογών. Ο κόσμος πραγματικά χειροκρότησε όταν καταφτάναμε στα εκλογικά κέντρα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι λοιπόν που είχαμε την δυνατότητα να παρευρεθούμε εκεί. Επτά ήταν οι αντιπροσωπείες ε, βουλευτών. Ο Ρόμπερτ Νόιτερ είναι εδώ, ήταν και αυτός μαζί μας. Και μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα τα οποία παρατηρήσαμε ήταν και τα περιορισμένα. Κυρίως ε, στην Καμπάλα, την ε, πρωτεύουσα και στις γειτονικές Τζίντζα και στην Μασάκα, στην γειτονική πόλη. Εγώ ήμουν στην, πήγα στην Τζίντζα και εσείς πήγατε στη Μασάκα, μάλιστα. Μας είπαν λοιπόν ε, οι άνθρωποι ότι ήμασταν στο λάθος μέρος. Μας έλεγαν στην Ήπεθρο θα έπρεπε να πάμε, στην, ε, στα χωριά, στις πόλεις, τι να δείτε. Και αυτό ίσως είναι ένα μάθημα το οποίο θα πρέπει να το συγκρατήσουμε για το μέλλον. Ό,τι άλλο το τι γίνεται στην πρωτεύουσα, αλλά το τι γίνεται στα χωριά. Παρ' όλα αυτά, με το, όπως είπε και ο κ. Σκούκαν, ήταν εξαιρετική συνεργασία και επιβεβαιώσαμε το παραπάνω τα απορίσματα της μακροχρόνιας και μακροπρόθεσμης αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι η παρουσία μας πραγματικά εκτιμήθηκε και της δόθηκε μάλιστα μεγάλη δημοσιότητα στον τύπο. Η ανάλυση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ε, κάτι που έπαιξε ρόλο κλειδί και για την αντίληψη του κόσμου σχετικά με τις προεδρικές αυτές ε, και βουλευτικές αυτές εκλογές. Σε ό,τι αφορά τη δεσμεύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουγγάντα, ο κ. Κούκαν αναφέρθηκε ε, στο ότι ήταν οι τρίτες εκλογές με τη συμμετοχή πολλαπλών κομμάτων. Ο ίδιος ο Πρόεδρος μας ε, δήλωσε ότι είμαστε νέα δημοκρατία και έχουμε πολλά να μάθουμε ακόμα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν στις συστάσεις μας του 2006 του 2011 και για τρίτη φορά λοιπόν τώρα όταν θα καταρτήσουμε συστάσεις θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν στη χώρα προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός ικανοποίησης σε ό,τι αφορά τις δημοκρατικές εκλογές. Λυπούμαστε γιατί δεν ήταν πολλές οι συστάσεις του 2011 οι οποίες εφαρμόστηκαν. Αντιθέτως, το νομικό πλαίσιο περιόρισε τον χρόνο ψηφοφορίας, ε, περιόρισε την διάρκεια της περίοδου ε, προεκλογικής εκστρατείας σε ό,τι αφορά επίσης ε, την διαδικασία καταχώρησης των υποψηφίων. Δημιούργησε δε επίσης 52 νέες επί εκλογικές περιφερειές. Και το υψηλό κόστος της συμμετοχής στις εκλογές απέτρεψε πολλούς. Είδαμε πάρα πολλές ε, εκθέσεις και μελέτες που καταδεικνύουν πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν άμεσα προς, τους, ε, προς το εκλογικό κοινό, προς τους ντόπιου. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορούμε αυτό να το αποδείξουμε, αλλά είχαμε στο ότι πρόκειται και για δημόσιους πόρους που ξόδεψε το κυβερνόν κόμμα στην προεκλογική εκστρατεία. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο αναφέρθηκε και το οποίο με εντυπωσίασε και εμένα σε ό,τι αφορά τη δημόσια τηλεόραση στις ειδήσει ο προεδρικός ε, ε, υποψήφιος είχε 11 ώρες στη διάθεσή του ενώ ο βασικός του αντίπαλος είχε τέσσερα λεπτά στη διάθεσή του σε, στις ειδήσεις σε ώρες αχμής. Αυτό σε ό,τι αφορά τη επικοινωνία στη χώρα αυτή, σε ό,τι αφορά το ραδιόφωνο, την τηλεόραση. Εδώ λοιπόν υπάρχει δυσαναλογία. 11 ώρες έναντι 4 λεπτών για τον βασικό υποψηφίο της αντιπολίτευσης. Να μην επαναλάβω αυτά που είπε ο κύριος Κούκα, να, να πω ότι σε ό,τι αφορά την τελική έκθεση θα δούμε πολλά, πολλές από τις συστάσεις μας να επαναλαμβάνονται, γιατί υπάρχουν ακόμα ελλείμματα. Η Ουγγάντα είναι ζωντανή χώρα, εξαιρετικοί, εξαιρετικοί άνθρωποι, νέοι άνθρωποι και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στο τμήμα αυτό της Αφρικής Άκουσα κάτι πολύ καλό, ότι πολλοί πρόσφυγες από τη Σομαλία, το Νοτιό Σουδάν, το Μπουρούντι, το Κονγκό, το Τσάντ βρίσκονται στην Ουγγάντα και δεν υπάρχουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα πολύ θετικό παράδειγμα. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν πάρει και ένα κομμάτι γης, έχουν δώσει για να μπορούν να στραφούν και να τρέψουν την οικογένειά τους. Πέρα λοιπόν από την κριτική που ασκούμε, θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά και τη νέα Επιτροπή Παρακολούθησης των Εκλογών θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με την κοινωνία των πολιτών για να βελτιωθούν οι όροι. Ευχαριστώ πολύ. Να πω απλώς ότι στα πλαίσια της ε, ενίσχυσης ε, της δημοκρατίας της πρωτοβουλίας. Προσπαθούμε και μεταξύ των εκλογών να παρέχουμε στήριξη και, δέσμευση και παρακολούθηση και όχι μόνο με τις αποστολές. Ε, δεν ξέρω αν η κυρία ε, Πρέσβης θα ήθελε να μας πει κάτι. Έχουμε μια δήλωση, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω εδώ τον αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου δίπλα μου, ο οποίος ε, θα κάνει μια δήλωση εκ μέρους της ε, αντιπροσωπείας της Ουγκάντα. Ναι, ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, μου είχαν πει ότι θα προσέλθει, μετά μου είπαν ότι δεν μπορούσε, τελικώς ζητώ συγγνώμη. Πάντως έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να συμμετέχουμε στην συζήτηση αυτή και στην συζήτηση με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να πω ότι πέρυσι ε, ε, εδέχθη μία αντιπροσωπεία στο γραφείο μου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με κάναμε μία προκατακτική μελέτη για να δούμε κατά πόσο ήταν απαραίτητο να έχουμε αποστολή παρακολούθησης ε, εκλογών. Είπαμε ότι εκφράσατε κάποιες υποψίες για τα όσα συμβαίνουν στην Ουγκάντα. Η προκαταρτική μελέτη λέγει ότι η νομοθεσία δεν ακολουθείται επαρκώς και άλλα και αυτό θα ήταν επαρκής λόγος για να πραγματοποιηθεί η αποστολή και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που έλαβε χώρα η αποστολή αυτή γιατί αν δεν είχε γίνει αυτή η αποστολή δεν θα διαξήγεται και αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή. Απεστάλλει λοιπόν η αποστολή αυτή στην Ουγκάντα. Είδαν οι συμμετέχοντες τα τεκτενόμενα στη χώρα. Υπευλήθησαν εκθέσεις σύμφωνα με αυτά που συζητούμε αυτή τη στιγμή. Προφανώς και χαιρετίζει το διάλογο η Δημοκρατία της Ουγκάντα, το διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα κοινού συμφέροντος. Για τα σημεία της εκθέσεως θα θέλαμε τα εξή να πούμε. Η, εκλογή, η Επιτροπή Εκλογών της χώρας κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να, επιτρέψει τη συμμετοχή στις εκλογές Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Και ως νεαρή δημοκρατία η Ουγγάντα αναπτύσσει τους θεσμούς της και τους ενισχύει. Έχουμε διέλθει μια διαδικασία μετα... εκλογικής μεταρρύθμισης για να βελτιώσουμε το δημοκρατικό σύστημα. Αλλά είχαμε και τροποποιήσεις και τροπολογίες. Είχαμε μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν και στην ε, εκλογή των μελών του Κοινοβουλίου και την μεταρρύθμιση του συντάγματος. Είχαμε συγκεκριμένο κύκλο μεταρρυθμίσεων το 1995, μετά το 2001 είχαμε εκλογές, μετά από άλλες μεταρρυθμίσεις το 2000, το ίδιο είχαμε και το 2005 και τότε ήμουν πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής των Μεταρρυθμίσεων, τότε ήταν το 2005. Το 10 είχαμε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στα εκλογικά θέματα και σύμφωνα με αυτές τις μεταρρυθμίσεις διεξήχθησαν αυτές τις τελευταίες εκλογές. Και εγώ ως αναπληρωτής πρόεδρος τότε παρακολούθησα τη διαδικασία αυτή μεταρρυθμίσεων και βελτιώσεων. Κάθε φορά που διεξάγονται εκλογές ανακαλύπτουμε κάποια κενά που πρέπει να καλύπτουμε μέσω μεταρρυθμίσεως. Αυτή η διαδικασία ήταν συνεχόμενη και γι' αυτό μας εκπλήσει κάπως ότι πέρυσι είχαμε εξωθήσει, είχαμε κάνει μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τις εκλογικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό το κάνουμε τακτικά, συστηματικά στην Ουγγάντα και επομένως δεν κατανοήσαμε γιατί ισχύει το αυτή η πίεση εκείνη τη στιγμή και αναπτύσσεται το πίεση και εκεί που δεν θα έπρεπε να υπάρχει οι εκλογικέ μεταρρυθμίσει, ε, τουλάχιστον στη δική μου εμπειρία, ήταν ότι όπω σα είπα, οι διαδικασίε αυτέ μεταρρύθμιση ήταν τακτικέ και συστηματικέ. Είμαι βέβαιο ότι αυτή τη συστηματικότητα την υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2005 θα θυμάστε, μάλλον θα θυμάστε ότι τον Ιούλιο του 2005 είχαμε το λεγόμενο πολιτικό σύστημα κινημάτων και μέσω δημοψηφίσματος το 2005 εγκρίναμε την, ε, το πολυκομματικό σύστημα ώστε να βελτιωθεί η δημοκρατική παράδοση στη χώρα. Είχαμε διάλογο με ομάδες ε, ενδιαφερόντων που μας είπαν ότι δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε έτσι. Θα έπρεπε να πάμε σε πολυκομματικό σύστημα και συζητήσαμε με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς για την ε, μεταρρύθμιση των εκλογών ή στο Σύνταγμα υπάρχει ένα διακομματικό φόρουμ, προβλέπει το Σύνταγμα, όπου όλα τα κόμματα συναντώνται και συζητούν για το τι θα πρέπει να συμβαίνει. Υπάρχει ένα κεντρικό γραφείο και όλες οι σημαίες των κομμάτων ανεμίζουν έξω από την πόρτα του κτηρίου αυτού. Ο διάλογος αυτός συνεχίζεται λοιπόν και η τελευταία μεταρρύθμιση ήταν πέρυσι σχετικά με την προεδρική εκλογή. Τροποποιήθηκε ο σχετικός νόμος όπως και ο νόμο, η νομοθεσία για την τοπική εκπροσώπηση βάσει της οποίας δηλαδή γίνονται οι τοπικές εκλογές η συμμετοχή, τα, οι ποσοστώσεις δηλαδή ανθρώπων με αναπηρία η εκπροσώπηση των φύλων ώστε να μπορούμε να υποβάλουμε ένα νόμο πλαίσιο για τη διευκόνηση των εκλογών. Το Φεβρουάριο του 2016, σύμφωνα με την ε, νομοθεσία τους, ε, την τροποποιημένη νομοθεσία, διεξήχθησαν και ε, ήταν ειρηνικές και δίκαιες. Τώρα υπήρχαν κάποια οργανωτικά προβλήματα που δεν είχαμε προβλέψει, δηλαδή η παράδοση των ψηφοδελτίων και η προμήθεια των ψηφοδελτίων, η ίδια η εκλογική επιτροπή ε, ε, έλαβε με πολύ μάλλον πολύ καθυστερημένα την ειδοποίηση για, ε, για τα προβλήματα αυτά της καθυστέρησης δηλαδή παράδοση των ψηφοδελτίων για το οποίο μάλιστα εξέδωσε και δημόσια συγνώμη εκεί όπου είχαμε κάποια προβλήματα επεκτάθηκε το, η προθεσμία κατά περισσότερο από δύο ώρες για να μπορέσουν να διεξαχθούν οι εκλογές. Μάλιστα σε κάποιες περιφέρειες προχώρησαν οι εκλογές μέχρι και την επόμενη μέρα. Μέχρι και τις 9 του περασμένου μήνα έγινε η προέκταση αυτή για κάποιες συγκεκριμένες περιφέρειες, 9 Μαρτίου. Οι εκπρόσωποι της ΟΑΚΑ μόνον την περασμένη Παρασκευή εξελέγησαν. Πρόκειται λοιπόν για μια δικασία που τρέχει ακόμη και εμείς την παρακολουθούμε και είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με τα όσα ε, συμβαίνουν και με τον τρόπο που διεξάγονται. Ο πρόεδρος Σεβένη του NRM ήταν ο νικητής των εκλογών 60,7% έλαβε 35,37% έλαβε το επόμενο κόμμα και μετά είχαμε τα ποσοστά που αναφέρατε κι εσείς. Μετά είχαμε την ε, αποστολή του Commonwealth, την αποστολή παρατήρηση του Commonwealth, για την επέκταση των, του ωραρίου της ε, προθεσμίας των εκλογών για να ασκηθούν τα δικαιώματα τα εκλογικά. Τώρα, πολλές από τις επικρίσεις που έγιναν είναι προς το δημοκρατικό συμφέρον της χώρας και η κυβέρνηση έχει καθήκον, έχει ευθύνη και καθήκον να προστατεύσει τον πληθυσμό, τους πολίτες της Ουγκάντα και την ιδιοκτησία τους. Δηλαδή, οποιασδήποτε ενδείξεις πληροφοριών θα έδειχναν μια προσπάθεια παρέμβαση στην ειρηνική αυτή διαδικασία ότι προετοιμάζονταν βίες διαδηλώσεις ή χρησιμοποίηση των ε, κοινωνικών φόρουμ ή άλλων για να διαταράξουν τη διαδικασία είχαν συμβεί και σε γειτονικέ χώρες πριν από κάποια χρόνια αυτά για να υπάρξει κινητοποίηση για βίες διαδηλώσεις ή βίες δράσεις και ορισμένα μέτρα ανελήφθησαν προς την προστασία του πληθυσμού μεταξύ των οποίων τα αναφέρατε και εσείς, τα μέσα κοινωνικών δικτύων μπλοκαρίστηκαν σε κάποιες περιοχές, περιορισμοί που επέτρεπε εν πάση περιπτώσει η νομοθεσία ανελήφθησαν προκειμένου να προστατευθεί ο λαός της Ουγκάντα και η διοκτησία του επί τη βάση των πληροφοριών που είχαμε εάν δεν ελέγχαμε ορισμένα, ορισμένες ε, κινητοποίησεις. Αυτό αφορούσε και τα ηλεκτρονικά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά έγιναν σύμφωνα με το του μήμα 31 της ε, νομοθεσίας για τις τηλεπικοινωνίες του 2013 σύμφωνα με, το, με τον έλεγχο του, του περιεχομένου των ηλεκτρονικών αυτών υπηρεσιών και την ε, κλίση σε βίες δραστηριότητες που προβλέπει η νομοθεσία εκείνη. Εμείς έχουμε απόλυτη ελευθερία και προστασία του τύπου και αυτό το εγγυάται το Σύνταγμα, αν δείτε το Σύνταγμά μας, όλες οι διατάξεις αυτές είναι εκεί. Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η προστασία της ελευθερίας του τύπου, η πρόσβαση των πολιτών ή στην ενημέρωση, οι αστυνομικές δυνάμεις είναι υπεύθυνε για την επιβολή του νόμου, για την προστασία της ιδιοκτησίας και για την διατήρηση της ε, ειρήνης. οι ειδικέ δυνάμεις ε, αποτροπής της αστυνομίας έχουν βελτιωθεί και έχουν κερδίσει και σε διαφάνεια, αλλά είναι απόλυτο μέρος και της ε, κοινοτική ειρήνευσης και επιβολής του νόμου, που από το 1999 έχει γίνει πολύ δημοφιλές και μεταξύ των πολιτών. Παρότι μπορεί κάποιες φορές να έχουμε δημοσιεύματα τα οποία δεν αποτυπώνουν πολύ ακριβώς τα πράγματα η αποτροπή του εγκλήματος, η σχετική μονάδα της αστυνομίας δεν είναι κάποιο, κάποια ένοπλη ε, μιλίσσα. είναι τμήμα της επίσημης ε, αστυνομίας της Ουγκάντα. Έχει σαφές νομικό πλαίσιο και η κυβέρνηση προετοίμασε ένα μνημόνιο έγκρισης πολιτικής και σχετικού σχεδίου νόμου για να χρησιμοποιούνται εθελοντές που ήταν αθρώοι. Είχαμε αθρώα προσέλευση εθελοντική προς το τμήμα αυτό της αστυνομίας. Που πολλοί πολίτες ήθελαν δηλαδή εθελοντικά να συμμετάσχουν στον μηχανισμό αποτροπής του εγκλήματος. Και γι' αυτό είχαμε όλους αυτούς τους αριθμούς των ανθρώπων και νεαρών που αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι αλλά που αντιλαμβάνονται ότι η κοινότητά τους, η τοπική τους κοινότητα θα πρέπει να ηγηθεί για την προστασία αυτή. Επομένως το αστυνομικό σώμα δρά απολύτως εντός του νομικού πλαισίου ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται ακραίες προκλήσεις από κάποιους. Και θα είδατε και εσείς στην Ουγγάντα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικές δυνάμεις και τον αυτοέλεγχο και την συγκράτηση που επέδειξαν έναντι των έντονων αυτών προκλήσεων. Και οι αστυνομικές δυνάμεις δεν παρενοχλούν δημοσιογράφους σε καμία περίπτωση. Ε, υπευλήθη, ε, υπευλήθησαν κάποια στοιχεία για ένα συγκεκριμένο κρούσμα, το εξετάσαμε πολύ σοβαρά δεν, ήταν όμως, ε, δεν πρόκειται όμως για μέλη ε, του αστυνομικού σώματος, σε καμία περίπτωση, οι οποίοι είχαν ελεγχθεί αυστηρά και συστηματικά καθ' όλη τη διαδικασία και μετά τις εκλογές. Μόνο όταν ενεργοποιείται το νομοσχέδιο ε, της... Όταν ενεργοποιείται το ειδικό νομοδιάταγμα της ε, δημόσιας τάξεως, τότε μόνον παρεμβαίνει η αστυνομία για τέτοιου είδους ε, διαδικασίες αποτροπές, αποτροπής και δίδονται και οδηγίες για την κυκλοφορία, για παράδειγμα, των οχημάτων. Πολλά καταστήματα αναγκάζονται να κλείσουν διότι περνάνε συγκεκριμένες πομπές ε, οχημάτων μπροστά ή μέσω τέλο πάντων βασικών αρτηριών. Η, η εκλογική επιτροπή είναι ένα απολύτως συνταγματικά εγκεκριμένο σώμα και τα μέλη της ορίζονται από τον πρόεδρο με την έγκριση του Κοινοβουλίου και ασκεί την ανεξαρτησία της η εκλογική επιτροπή για παράδειγμα Ε, συγκεκριμένος υποψήφιος για την προεδρική εκλογή συμπεριελήφθη στον κατάλογο παρά, το γεγονός ότι κρατείτο σε φυλακή υψής της ασφαλείας. Η ναψένσα όμως η εκλογική επιτροπή με αντίστροφη γνωμοδότηση της κυβερνήσεως τον, τον ε, συμπεριέλαβε στον κατάλογο των υποψηφίων. Και όπως λέγει και η παρατήρηση εκλογών της Ανατολικής Αφρικής, η διαδικασία των εκλογών έχει αποκεντροποιηθεί και αυτό ενισχύει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας για την ε, καταμέτρηση των ψηφοδελτίων ε, το ευρύ κοινό ήταν μάρτυρας της διαφανής διαδικασίας εδόθη αντίγραφο το οποίο είχε αναρτηθεί σε εμφανές σημείο σε κάθε εκλογικό κέντρο τα εκλογικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν και τοπικά και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής και δίνουν τα ακριβή αποτελέσματα αναδιαμέρισμα και αναεκλογικό κέντρο και μέχρι σήμερα είναι πολύ σημαντικό φόρουμ ενημέρωσης, η ιστοσελίδα της Επιτροπής, ε, για την έγκαιρη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και νεωτέρων για τις εκλογές. Και μέσω της τεχνολογίας βελτιώσαμε και την διαφάνεια του συστήματος, όπως και για την ταυτοποίηση των ε, ψηφοφόρων, χρησιμοποίησαμε ηλεκτρονικά συστήματα για να έχουμε και τα έγκαιρα, την έγκαιρη καταμέτρηση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων εντό οκτώ ώρων από τι εκλογέ, όπω προβλέπει η νομοθεσία. Όλα αυτά τα παρέχει ένα αναλυτικότατο νομοθετικό σχέδιο. Η διοικητική αρχή κάνει τις απαραίτητες ε, προετοιμασίες για την οποιαδήποτε επίλυση διαφορών με συγκεκριμένα καταρτισμένους ε, ε, δικαστικούς και δήλωσε ότι ήταν ικανοποιημένη με, την, το επίπεδο προετοιμασίας της. Οποιαδήποτε διαφορά υποβληθεί αυτή τη στιγμή μπορεί να προσφεύγει στα δικαστήρια. Οποιαδήποτε προσφυγή εξετάζεται εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπει ο νόμος. Και τα δικαστήρια της χώρας θα επικυρώσουν το κατά πόσον η εκλογική διαδικασία τελικά αποτυπώνει τη βούληση του λαού. οποιαδήποτε καταγγελία σε σχέση με προσφυγή προς το δικαστήριο θα εξεταστεί σε κάθε περίπτωση το αστυνομικό σώμα δεν, είναι, δεν ενέχεται σε καμία από αυτές τις προσφυγές και αν έχει υπάρξει τέτοια ενημέρωση ή ένδειξη αυτό στρεβλώνει την εικόνα της χώρας. Εμείς χαιρετίζουμε πάντως τις ε, ε, εκλογικέ αποστολές και θεωρούμε ότι συνεισφέρουν στην καλύτερη συμμετοχή του λαού, του κόσμου. Και επειδή αναφερθήκατε για την, ε, για την ισότητα των φύλων, υπάρχουν διάφορα ζητήματα κοινωνικο-οικονομικά για την συμμετοχή των γυναικών. Αυτό, αυτά είναι κοινά προβλήματα σε όλο τον κόσμο για τις γυναίκες. ίσως να είναι ακόμα δυσχερέστερη ή δυσμενέστερη η κατάσταση στις πιο φτωχές χώρες, αλλά η Ουγγάντα οπωσδήποτε έχει καταστήσει προτεραιότητα την ισότητα των φίλων στην πολιτική μαζί με, τον, ε, με την οικονομία και τον δημόσιο τομέα. Η συμμετοχή μιας γυναίκας ε, στον κατάλογο των υποψηφίων προεδρών είναι ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση. Σας θυμίζω ότι σε αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες ακόμα και η έννοια της γυναίκας υποψηφίου είναι κάτι το πολύ μακρινό. Σχεδόν αδύνατο σε κάποιες χώρες. Αλλά είχαμε ενισχυμένη συμμετοχή των γυναικών και στην εκλογική διαδικασία και στην πολιτική διαδικασία. Στην Ουγκάντα η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική είναι κάτι προς το οποίο, ε, το οποίο μάλλον ένθερμα υποστηρίζει όλος ο λαός. Και θεωρούμε ότι θα διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Έχουν ανεβεί προσπάθειες για την συμμετοχή και την προστασία των ανθρώπων με αναπηρία και οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση είναι ακαλοδεχούμενη προς αυτήν την κατεύθυνση. Κλείνοντας θα ήθελα να επαναλάβω τη δέσμευση της ε, κυβέρνησης της Ουγκάντα να συνεχίσει το διάλογο με αυτοσεβασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Σας ευχαριστώ. Uh, uh, ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους που επιθυμούν ε, να πάρουν το λόγο. Να δώσω καταρχάς το λόγο στον κύριο Νόιζερ που ήταν μέλος της αποστολής. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ακούγοντα και την δήλωση τη αντιπροσωπεία από την Ουγγάντα, θα είχε κανεί την εντύπωση ότι όλα πήγαν καλά. Δεν ε, ισχύει αυτό, αλλά πολλά ήταν καλά. Και με την ε, επιτροπή μας, με την αποστολή μας, είδαμε ότι έχουν γίνει μεγάλη πρόοδοι και στη συνέντευξη τύπους και στις συζητήσει με τους ε, δημοσιογράφους, παράλληλα με την αποστολή παρατήρησης. Ακούσαμε αυτό το παράδειγμα του κατά πόσον ε, το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο και τελικά καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι σε κάθε περίπτωση το ποτήρι είναι μισογεμάτο. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι σε θετική εξέλιξη. Θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω το εξή. Ο συνάδελφος Κούκαν και ο συνάδελφος Γεωλάινεν έκανε εξαιρετική δουλειά σε ό,τι αφορά και την παρατήρηση από τον κύριο Κούκαν, θεωρώ ότι δημιούργησε μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ουγγάντα και είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους τρεις υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου και είχαμε και δύο ώρες με τον Μουσέβνη την ε, ημέρα πριν από τις εκλογές, το βράδυ πριν από τις εκλογές. Αφιέρωσε πραγματικά τόσο χρόνο στην ε, αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πραγματικά ήταν καλή η ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να μην ξεχάσω σε καμία περίπτωση και τους υπαλλήλους μας, οι οποίοι τα διοργάνωσαν όλα εξαιρετικά. Υπήρχαν και δύσκολα στιγμές άλλωστε. Επικράτησαν κάποιες μικρές ε, αναταραχές και ήταν πολύ σωστή η αντίδραση τη αντιπροσωπείας μας και πραγματικά είναι σημαντικό να υπάρχει εμπειρία σε τέτοια ζητήματα. Αναφέρθηκαν κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά το θέμα της, του ελέγχου των κοινωνικών μέσων και του μπλοκαρίσματος των κοινωνικών μέσων. σε ό,τι αφορά την, το ρόλο της ε, εκλογική επιτροπής. Εδώ πραγματικά είδαμε υπερβολικά μικρή εξέλιξη και μικρή πρόοδο σε σχέση με το 2006 και το 2011 και θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη ανεξαρτησία πραγματικά σε ό,τι αφορά την εκλογική επιτροπή αυτή στο μέλλον και να υπάρξει και μεγαλύτερη δέσμευση από ό,τι έως τώρα. Να διευκρινίσω ότι είχαμε διάφορα περιστατικά την ημέρα των εκλογών, ότι για παράδειγμα ε, τα ψηφοδέλτια που δεν ε, ήταν στη διάθεση του κόσμου για δύο ώρες και ο κόσμος παρόλα αυτά περίμενε δύο ώρες. Και στην Ευρώπη πραγματικά οποιαδήποτε εκλογική επιτροπή θα είχε εξαναγκαστεί σε παρέτηση μετά από τέτοια περιστατικά. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να γίνουν αλλαγές. κάπως έκπληκτοι και σοκαρισμένοι ήμασταν με το γεγονός ότι ο Μπεζίτσο, ο βασικός αντίπαλος του Προέδρου Μουζίβενη, στο διάστημα το σύντομο που βρεθήκαμε στη χώρα, ε, συνελήφθη τρεις φορές και συνοδεύτηκε στην οικία του, κατανοώ κάπως και την κυβέρνηση της Ουγκάντα, η οποία δήλωσε ότι ο Μπεζίτσο προέδισε σε προκλητικές ε, συμπεριφορές, αλλά εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπήρχε μεγαλύτερη κυριαρχία για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Κάτι άλλο πολύ θετικό και το σημειώνω είναι ότι το Σαββατοκυριακό πριν την ημέρα των εκλογών έγινε μια συνομιλία μεταξύ των υποψηφίων την οποία δεν έχω ξαναζήσει τέσσερις ώρες live με αναμετάδοση συζήτηση με τους οκτώ υποψηφίους και αυτό αποτελεί μια σαφή ένδειξη για τη στάση της Ουγκάντα. Αυτό το καταδεικνύουν και τα σύμβολα, τα σύμβολα τα οποία τα επισημαίνουμε. Όταν λοιπόν οι οκτώ υποψήφοι πριν από τις εκλογές ε, ανταλλάσσουν χειραψίες και μαζί τραγουδούν τον εθνικό ύμνο και προσεύχονται, αυτό νομίζω ότι καταδεικνύει αξιοσημείωτε εξελίξει στην Ουγγάντα. Τέτοια λοιπόν σημαντικά σύμβολα δείχνουν ότι η Ουγγάντα είναι στο σωστό δρόμο. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι εκτιμούμε ιδιαίτερο τη στάση και την εξέλιξη της Ουγγάντα. Μετά από τον εμφύλιο έχει εξελιχθεί σε μια σταθερή δύναμη στη γενικότερη περιοχή. Και ασφαλώς και θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρατρύνουμε τη διαδικασία αυτή. Κοιτώντα ε, τη δημοκρατική εξέλιξη, το ίμιση των κατοίκων τη Ουγγάντα δεν μπορούσε καν να ψηφίσει γιατί ήταν κάτω των 18 ετών. Βλέπουμε λοιπόν ποιες είναι οι προοπτικές για την χώρα. Και εδώ θα πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο θέμα είναι η συνεργασία με τους ΜΚΙΟ. Θα πρέπει και αυτή να συνεχιστεί. Και αυτό θα ωφελούσε, θεωρώ, τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Συνολικά, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι οι εκλογές ανέδειξαν σαφή νικητή. Η χώρα έμεινε σχετικά ήσυχη και ήρεμη. Και προσβλέπουμε στην ε, μελλοντική συνέχιση της συνεργασίας με την Ουγκάντα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, Νόρμπερτ. Να πάσω τώρα το λόγο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τον κύριο Στεφανάρης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις που ακούσαμε, για τις ομιλίες για τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και να συγχαρώ πρώτα απ' όλα τον κύριο Κούκαν που ήταν επικεφαλής των παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γιώ Λέινεν, τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας. Σίγουρα η συνεργασία και με τον πρόεδρο της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν πάρα πολύ καλή. Η παρατήρηση λοιπόν ξεκίνησε το Δεκέμβριο και θα μείνει μέχρι την ε, κατάληξη της απόφασης στον νότο του δικαστηρίου όσον αφορά την προεκλογική διαδικασία και τις εκλογές. Είναι εμφανής η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη δημοκρατία στην Ουκάντα τα λέμε αυτά και στην προκαταρκτική μας έκθεση και λέμε και τα προβλήματα που υπήρχαν, εκφοβισμός, ε, στον αφορά φωτογραφίες, περιορισμό στα μέσα ενημέρωσης των πόρων προς τους υποψήφιους, ότι δεν υπήρχε ανεξαρτησία στην ε, εκλογική επιτροπή και καθυστέρηση των ψηφοδελτίων στα εκλογικά κέντρα, κάτι το οποίο οδήγησε ε, στο να ψηφίσουν λιγότεροι από όσοι κανονικά μπορούσαν να ψηφίσουν στις εκλογές αυτές. Όλες αυτές οι ανησυχίες πρέπει να καθισχαστούν. Επίσης, μας απασχόλησε πολύ και η ιδέα της αστυνομίας. Και οι δυσκολίες που αντιμετώπισε η αντιπολίτευση, που πήρε 35% και τσοπεζή και σύμφωνα με την Επιτροπή Εκλογών. Δεν υπάρχει καμία ε, καταγγελία κατά του Πεζίκε, ο οποίος όμως κρατείται παρόλα αυτά. Το άλλο που ζητάμε είναι όλες οι πλευρές να αποφύγουν οποιαδήποτε πράξη ή δράση που θα ανακαινούσε βία στη χώρα. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής της Ουγκάντα βρίσκεται εδώ σήμερα και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό που μπόρεσε να ακούσει και την παρουσίαση του κύριου Κόκαν. Σας ευχαριστούμε και εσάς για τόσα είπατε. Η παρουσία σας εδώ δείχνει τη σημασία που δίνει η Ουγκάντα στη συνεργασία μας σε μια εταιρική σχέση που υποστηρίζει τη δημοκρατία. Συνεχίζουμε τη συνεργασία μαζί σας με τις αρχές της Ουγκάντα. Τα αποτελέσματα των ε, παρατηρητών, τα συμπεράσματά τους, ε, καταλήγουν στο ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος στην εκλογική διαδικασία. Εμείς από τη δικιά μας την υπηρεσία προσβλέπουμε στην τελική έκθεση η οποία θα συμπεριλαμβάνει και συστάσεις για τους διάφορους παράγοντες που εμπλέκονται στις εκλογές αυτές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία έχει να προσθέσει τίποτα. Όχι. Καλώς. Πρόκειται για τις εκλογές εξάλλου, όντως. Κύριε Κούκαν, θέλετε να απαντήσετε σε κάτι από αυτά που ακούσατε, είτε στον ομιλητή μας από την Ουγκάντα, είτε σε κάποιον άλλον, ο κύριος Κούκαν. Ναι, να αντιδράσω κάπως σύντομα. Δύο-τρεις παρατηρήσεις για να έχουμε τη συνολική εικόνα. Δεν ανέφερα πριν τον ενεργό ρόλο της Σουγκάντα στην περιοχή. Είναι κάτι που εκτιμούμε όλος ιδιαίτερος. Έχει πολύ θετικό ρόλο υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, αν λάβουμε υπόψη μας στο Σουδάν, τη Σομαλία που βρίσκονται εκεί, έχει διαμεσολαβήσει η Ουγκάντα, Μπουρούντι και εκεί. Και αυτό πρέπει να το πούμε και να το υπογραμμίσουμε. Θέλω επίσης να αναφέρω και τότε υπάρχουν πολλοί διεθνείς παρατηρητές στην Ουγκάντα. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά μεταξύ μας. Είχαμε συναντήσεις, εντάξει δεν σκοπεύαμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό ανακοινοθέν γιατί προφανώ η οπτική μας γονείται διαφορετική αλλά η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι ένα καλό νέο στοιχείο στο όλο αυτό πλαίσιο παρατήρησης των εκλογών. Εκτιμούμε όλους ιδιαίτερως λοιπόν το ρόλο της Ουκάντα και άκουσα προσεκτικά το είπατε κι εσείς. Κατάλαβα πολλά από αυτά που αναφέρατε. Υπάρχουν μερικά σημαντικά ζητήματα από τη δική μας την πλευρά που δεν αναφέρατε και μπορώ να καταλάβω γιατί. Εγώ αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες σας όσον αφορά την ασφάλεια. Αλλά δεν εξηγούνται όλα επειδή κάποιος ανησυχεί για την ασφάλεια. Ιδίω όταν τα επιχειρήματα αυτά θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τις μυστικές υπηρεσίες. Αυτό που κυρίως εκτίμησα στα όσα μας είπατε είναι η επαναλαμβανόμενη δέσμευσή σας για διάλογο ουσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το καλασαρίζω αυτό, γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουγκάντα είναι τέρος. Θέλουμε να έχουμε ισχυρές σχέσεις μεταξύ μας. Και γι' αυτό πρέπει να μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά μεταξύ μας για όλα τα ζητήματα. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε θέσεις που θα βοηθήσουν την Ουγκάντα και το λαό της. Οπότε προσβλέπω στη συνέχιση του διαλόγου αυτού. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ όλους. Όντως, η εταιρική αυτή σχέση με την Ουγκάντα είναι σημαντική για μας και η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών εκεί. Η δημοκρατία προσφέρει καλύτερη ζωή στους λαούς μας και σε αυτό προσβλέπουμε. Οπότε θέλουμε και στο μέλλον να συνεργαστούμε μαζί σας προς αυτή την κατεύθυνση. Και ελπίζω να έχουμε παρετέρω συνεργασία και στο μέλλον μαζί για όλα αυτά τα θέματα που θίξαμε εδώ. Ωραία συνάδελφοι, καλώς. Τελευταίο θέμα μας, το σημείο 11. Αλλιευτικές δυνατότητες με την Μαυριτανία. Εδώ θα είμαστε πιο σύντομοι, γιατί νομίζω ότι δεχόμαστε τις συστάσεις, να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας δηλαδή σε αυτό. Ο Εγνάθιο Καράου έχει το λόγο που είναι ο συντάκτης γνωμοδότησης. Παρακαλώ. όπως έλεγε η πρόεδρος, μια σύντομη έκθεση στην οποία μπορούσαμε να πούμε απλώς ναι ή όχι. Αυτό που δεν με ικανοποιεί είναι περισσότερο το γεγονό ότι δεν είμαστε πλέον πολύ στην αίθουσα παρότι επαναλαμβάνω δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε την συμφωνία αυτή παρά μόνο να συνενέσουμε ή όχι ε, θα ήθελα λίγο, θα με ενδιαφέρει να συζητήσουμε πώς λειτουργούν αυτές οι εκθέσεις της ΔΕΒΕ, αλλά και πώς λειτουργεί συνολικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στο πλαίσιο των συμφωνιών. Διότι αλλιώς εκκρεμόμαστε από αυτό το άρθρο 99 που εισήχθη στον κανονισμό για να πούμε ναι ή όχι. Δηλαδή, αν θέλετε, υπάρχει ένα πρόβλημα ε, δημοκρατικού ελέγχου απέναντι σε αυτά που μας προτείνει η Κομισιόν. Επιπλέον μιλούμε εδώ για την Μαυριτανία που είναι, έχει διάφορα προβλήματα, είναι μια φτωχή χώρα και για την οποία οι αλληλευτικές συμφωνίες είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Επί της ουσίας τώρα εδώ δεν μπορούμε όμως να τοποθετηθούμε παραπάνω να, όπως έλεγα, να συνενέσουμε ή όχι. Θα ήταν χρήσιμο, θα ήταν καλό αυτή η Επιτροπή να παρέμβει παρόλα αυτά επί της ουσίας της συμφωνίας, της προτάσεως δηλαδή. Γιατί είναι μια σημαντική χώρα η Μαυριτανία που είναι και αναπτυσσόμενη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το θέσει αυτό η πρόεδρος ή στην συνάντηση των ε, πρόεδρων. Δηλαδή να θίξει την όλη προβληματική της χρησιμοποίηση της διατάξεως του άρθρου αυτού και ίσως μέσω του άρθρου 53 να συζητήσουμε αυτά περιεχόμενα των συμφωνιών αυτών των αλλιευτικών και στην Επιτροπή Ελίας. Γιατί και αυτοί δεσμεύονται με τον ίδιο τρόπο. Είτε συνενούν, είτε δεν συνενούν και τίποτε άλλο. Δηλαδή, για το περιεχόμενο εμείς θα εκφραζόμασταν θετικά, καταφατικά. Αλλά διαδικαστικώς πώς νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε. Ναι, ευχαριστώ λέει Γνωρίζω ότι έτσι λειτουργεί αυτή η διαδικασία μόνο με απλή συνένεση ή όχι και δεν μπορούμε να έχουμε προϋποθέσεις προκειμένου να συνενέσουμε αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιρροή του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, για παράδειγμα, η, αντίστοιχο, η αντίστοιχη θέση μας ως προς την TTIP δεν μας έχει υποχρεώσει, δεν μας έχει περιορίσει στην επιρροή που προσπαθούμε να ασκήσουμε. Μπορούμε να καλέσουμε την Κομισιόν να έρθει να μας τα εξηγήσει αυτά. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε σε γρήγορη επιταχυμένη διαδικασία. Μπορούμε να πάρουμε το χρόνο μας. Υπάρχουν πολλές ε, διαπραγματεύσεις εντός των οποίων μπορούμε να ασκήσουμε μια κοινοβουλευτική πίεση και επιρροή, παρότι στο τέλος η νομοθεσία πράγματι προβλέπει συνένεση ή όχι, ναι ή όχι το οποίο νόμος ε, και δεν συμπεριλαμβάνει δηλαδή ε, επί της ουσίας ε, προτάσεις για το τι θα έπρεπε να περιέχει. Επαναλαμβάνω ότι και στην TTIP ναι ή όχι έχουμε στο τέλος, αλλά έχουμε δαπανίσει αρκετό χρόνο και προσπάθεια εκεί. Είναι ένα κοινό πρόβλημα δηλαδή, έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα δεν βλέπω κάποιον συνάδελφο να ζητάει το λόγο επ' αυτού. Δεν ξέρω αν η DG είναι εδώ. Θέλετε κάτι να σχολιάσετε ε, για τη Μαυριτανία. Μήπως θέλετε εσείς ε, να υποβάλλετε κάποια ερώτημα στην Κομισιόν, στην DG Mare. Αυτό που έλεγα είναι ότι θα ήταν καλύτερα να το συζητήσουμε στην Επιτροπή αντί να απλώς να πούμε ναι ή όχι αυτό τη λειτουργία και έχετε δίκιο. Και στην TTIP το ίδιο ισχύει, δεν είναι καλό και εκεί. Ναι, η CFP μόλις μεταρρυθμίστηκε, δεν ξέρω αν θα το ξανανοίξουμε το θέμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξε μια, μια ριζική μεταρρύθμιση όλων αυτών του, του πλαισίου δηλαδή των αλλιευτικών συμφωνιών και αυτή εδώ είναι ίδια με άλλε ως προς το περιεχόμενό της. Όμως είναι χρήσιμο να μπορούμε να συζητούμε συγκεκριμένα ζητήματα με την, Κομισιόν, με την Κομισιόν. Μπορούμε να του καλούμε να συνομιλούν με τους ε, εισηγητέ και αν κάποιο δεν έχει ικανοποιηθεί, αυτό είναι το κατάλληλο βήμα. Η Κομισιόν είναι εδώ για να απαντήσει στα ερωτήματά μα. Δεν ξέρω λοιπόν αν η ΜΑΡΕ θέλει να μα πει κάτι για τη Συμφωνία τη Μαριτανία ή αν κάτι επέφεραν οι μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνει το λόγο, τον παίρνω ευχαρίστω, δεν θα μακρηγορήσω, αλλά θα ήθελα να διαφημίσω δύο πράγματα για τη συμφωνία αυτή. Και βεβαίω δεν πρόκειται να σχολιάσω τι ε, διαδικασίε υπό την νομοθεσία. Όπω είπε και η Πρόεδρο, εμεί σεβόμαστε τη συνθήκη και απλά εφαρμόζουμε τι διατάξει τη. Τώρα, για την συγκεκριμένη συμφωνία είμαστε θέση σα βεβαίω και σε οποιοδήποτε βήμα ή φόρμα να συζητήσουμε και το κάνουμε και στην Επιτροπή Αλίας, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και για άλλες επιτροπές. Είμαστε στη διάθεσή σας, επαναλαμβάνω. Και διμερός δηλαδή και με όποια άλλη μορφή θέλετε να το συζητήσουμε. Τώρα, εφόσον μου δίνετε κάποιο λεπτό, απλώς να πω ότι είναι ουσιώδης ε, αλλιευτική συμφωνία αυτή, είναι η πρώτη που έχουμε 55 εκατομμύρια ευρώ ε, είναι σημαντικός ο φάκελος για το πλαίσιό του, ε, αφορά και σημαντικό τμήμα του στόλου του Εωραϊκού, αρκετά ήδη και πάνω των 10 κρατών μελών της Εωραϊκή Ένωσης πρόκειται για μια ουσιαστικότατη συμφωνία και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ανανεώσαμε τις διαπραγματεύσεις με την Μαυριτανία διότι είχαμε πάρα πολλές διακοπές, για να το πω έτσι, πέρυσι από την υπογραφή τον περασμένο Νοέμβριο ε, μπορέσουμε να επανέλθουμε στις συνομιλίες ε, στην ε, κοινή χρήση της ελευτικής ζώνης Μαριτανίας και ιδιαίτερα δύο στοιχεία έχουν σημασία εδώ είναι η βιωσιμότητα των πόρων ήμασταν εξαιρετικά προσεκτικοί για να μπορέσουμε να αποδεχθούμε ελευτικές δυνατότητες μόνο επί των ειδών για τα οποία είχαμε συγκεκριμένες επιστημονικές αποδείξεις ότι έχουμε απόθεμα. Υπήρχαν ήδη κεφαλοπόδωνα, για παράδειγμα, που δεν απεδέχθημεν. Έχουμε ποσοστώσεις και κουότα για τα απελαγικά. Επίσης ε, ουσιαστικό στοιχείο του πρωτοκόλου για τις ε, σαρδέλες, ε, το σκουμπρί και άλλα από 300.000 τόνους προηγουμένως ε, περάσαμε στους 247 αν ακούσαμε καλά. Επομένως και εδώ έχουμε συγκεκριμένη επιφύλαξη και προσοχή για την παρακολούθηση των ειδών. Για είδη όπως ο, τόνος ε, μπορέσαμε αντιθέτως να αυξήσουμε σχετικά τις ποσότητες. Τώρα, ε, ανάλογα με την περίπτωση θα μπορέσουμε να επαναξετάσουμε για νέα είδη τις, ε, τις ε, δυνατότητες εφόσον οι επιστημονικές εκθέσεις μας το επιτρέψουν και εφόσον η Μαυριτανία μας διαθέσει ένα μέρος του αποθέματος. Τώρα, εδώ είναι χρήσιμο να θυμίσουμε ότι είχαμε σημαντική ε, διαφορά από το προηγούμενο πρωτόκολλο. Περάσαμε στα 55 εκατομμύρια ευρώ Δηλαδή είχαμε μία μείωση, λαμβάνοντα όμως υπόψη και την τροποποίηση και τη ευθυγράμμιση των αποθεμάτων των πόρων σύμφωνα με τις εκθέσεις. Είναι όμως πιο λογικό ε, αυτό το ύψο, αυτό το μέγεθος και αφορά και στην ε, αλλιευτική δραστηριότητα του οραϊκού στόλου. Τώρα για το αναπτυξιακό έχουμε μία στήριξη τομεακή για την καλύτερη διαχείριση του τομέα στη Μαυριτανία και στις ε, άλλες χώρες εταίρους για να μπορούμε να στηρίξουμε την τοπική αλληλεία, για να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα και την ανάπτυξη και να βοηθούμε την ανάπτυξη του κλάδου σε βιώσιμο πλαίσιο. Από 3 εκατομμύρια λοιπόν αυξήθηκε σε άνω των 4 η συνεισφορά μας αυτή, η ενίσχυση αυτή. Βεβαίως έχουμε μία σειρά προϋποθέσεων ε, για την χρηστή διαχείριση των πόρων αυτών και κριτήρια τα οποία πρέπει να γίνονται σεβαστά ε, και έχουμε και πρόσφατη έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου σχετικά με τη χρησιμοποίηση των πόρων αυτό που μας δεσμεύει. Αυτές λοιπόν οι βασικές αρχές που διέπουν την διαπραγμάτευση έχουμε τετραετή συμφωνία, το προηγούμενο πρωτόκολλο ήταν διετές. Έχουμε λοιπόν ένα σταθερό νομικό πλαίσιο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον κλάδο. Είχαμε διάφορες βελτιώσεις και υπό την τεχνική σκοπιά Έχουμε δύο διατάξεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες για την ε, αναπτυξιακή δυνατότητα της χώρας. Ε, είναι η καταρχάς χρησιμοποίηση στο 60% τοπικών ναυτικών. Τώρα έχουμε μια μικρή διαφορά για, για την βάση υπολογισμού αυτού του 60% αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα το επιλύσουμε στην Κοινή Επιτροπή πολύ γρήγορα για τα, είναι, στα τέλη Απριλίου θα είναι αυτό. Επίσης έχουμε υποχρεωτικές εκφορτώσεις στο 2% για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις ε, διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού αλλά και κάποια άλλα προβλήματα που έχουμε προσφύγων από, από το Σαχέλ. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά συνιστούν ένα θα έλεγα πολύ καλά ισορροπημένο πρωτόκολλο και βλέπω και μία σύστασή σας που λέει να έχουμε ευρύτατη συνένεση, ομοφωνία ενδεχομένως. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πρωτόκολλο αυτό. Ευχαριστούμε για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε για τη συμφωνία και για τις αλλαγές. Ωραία. Αύριο θα ψηφίσουμε. Αύριο. Έτσι έχει καθοριστεί και ίσως θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να βελτιώσουμε κάπως τη διαδικασία. Οι συντονιστές θα μπορούσαν να το συζητήσουν αυτό. Καλώ, σας ευχαριστώ πολύ όλους συνάδελφοι. Έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συνεδρίαση. Αύριο θα βρεθούμε και πάλι στις 9 για την ψηφοφορία, αρχίζοντας από την εμπορική συμφωνία. Και μετά θα ακούσουμε για τα άλλα θέματα, κλπ.